Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. La séance est ouverte. Να έχει συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, θεωρώ ότι η μερίσια διάταξη υιοθετείται. Δεν έχω καμία ανακοίνωση να σας κάνω. Και επομένως, θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Σας παρακαλώ, βάλτε τις τεχνικές σας κάρτες στις ε, συσκευές σας. Ας κάνουμε μια πρώτη δοκιμαστική ψηφοφορία. Έναξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. πρώτη ψηφοφορία. Είναι η έκθεση του κ. Γιάννη Σιγκέγερ για τον ΕΝΙΣΑ. Οργανισμός για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Πρόκειται για έναν κανονισμό, έτσι. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 14 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 3 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 16 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 5 υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείται. 18, 19 και 20 είναι οι ίδιες τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 17, καταπίπτει. 6, 7, υπέρ, 7 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε, 1 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε, 9 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 10 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε, 11 υπέρ, κατά, όχι, θα επαληθεύσουμε την 10. Ένα ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Καταπίπτει. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Θα την επαληθεύσουμε την 11. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας φοφορίας. Υιοθετείτε. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Υιοθετείτε 12 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε Και το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα. της ψηφοφορίας. Υιοθετείτε με 22 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα, για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για το σύνολο του κειμένου. Με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρσοφοριάς. Εγκρίνεται με 24 ψήφους κατά, 2 ψήφους, 24 ψήφους υπέρ, συγγνώμη, 2 ψήφους κατά. Ε, συγχαρητήρια και Φερνάντες για το σχέδιο διορθωτικού προ... προϋπολογισμού υπαριθμών 1 στο γενικό προϋπολογισμό του 18. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά. Τώρα, για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Είναι η έκθεση της κυρία Γκουαρδία Θαβάλ. Τεχνική βοήθεια. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4. Πρέπει να ψηφίσουμε δύο φορές εδώ. Για το πρώτο τμήμα του 4. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ναι, απορρίπτεται. Με 20 ψήφους κατά, 9 ψήφους υπέρ. Ήταν το δεύτερο τμήμα που απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται 7 υπέρ. Κατά. Άποχες. Υιοθετείται 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με 25 ψήφου υπέρ, 4 ψήφου κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Κύριε Γκουαρία θα Τώρα, για τη μεταφορά που προκύπτει από την προηγούμενη ψηφοφορία είναι μια ψηφοφορία που πρέπει να κάνουμε κατά συνέπεια της προηγούμενης, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα, παρακαλώ. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά. Τώρα, για τα άλλα τμήματα, για την τροποποίηση και το κείμενο του ελεγκτικού συνεδρίου. Ο εισηγητής δεν είναι παρόν, ο κ. Ashworth, τα υπόλοιπα τμήματα του προπολογισμού. Ίσως ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου είναι εδώ παρόν. Ίσως θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια για το θέμα αυτό. Αλλά δεν υπάρχουν ουσιαστικά επιπτώσεις στον προπολογισμό για τον, την προσαρμογή του προσωπικού. Δεν υπάρχει κανένας. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Βεβαίως, να σε εξηγήσω εγώ. Εκπροσωπείτε δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο. Βεβαίως, ναι. Πρόκειται για δύο αλλαγές που δεν έχουν δημοσιονομική επίπτωση. Δύο θέσεις, AST, ε, θα γίνουν AD. Ήταν θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Ε, μιλάμε για τη διεύθυνση πληροφορικής για τη μία θέση και κτηρίων, το άτομο αυτό θα είναι επιφορτισμένο με, το service desk και με τις υπηρεσίες και θα έχει και επίσης στην άλλη θέση μάλλον θα υπάρχει ένα άτομο μια διοικητική θέση με συντονιστικές αρμοδιότητες. Επίσης, θα έχει ε, αρμοδιότητες για την προστασία των δεδομένων. από τις 25 Μαΐου του 2018. Έχουμε μία θέση για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ένα άλλο για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων. Ε, υπάρχει ένα άτομο που θα, πάει στη σύνταξη, θα βγει στη σύνταξη από μια θέση AST και θα θέλαμε να προσλάβουμε ένα άτομο ε, AD ε, που γνωρίζει, έχει τεχνικές γνώσεις και θα αναλάβει τη θέση αυτή. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερε παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Η τροποποίηση του οργανογράμματος ε, μπορεί να υιοθετηθεί. Τώρα για την κτηριακή πολιτική δεν θα ψηφίσουμε και επομένως τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Και τώρα, θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας παρουσίασε στις 2 Μαΐου. Πρόταση για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος ήρθε στις 3 Μαΐου. Όλοι θα θυμούνται ότι δεσμεύτηκε να γίνουν οι εργασίες με την ομάδα του και τη γραμματεία μας, ούτως ώστε να διευκρινίσουμε κατά πόσο τα νούμερα είναι συγκρίσιμα. Δύσκολο είναι να κάνουμε συγκρίσεις δεδομένου του ότι τα προγράμματα αλλάζουν, είναι λιγότερα, υπάρχουν ομαδοποίησεις των προγραμμάτων και οι βάσεις λοιπόν σύγκρισης είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Αντίθετα με τη δέσμευση που είχε αναλάβει ο Επίτροπος, δεν κατέστη δυνατό να έρθουν σε επαφή δύο, οι δύο ομάδες και να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα δεδομένα. Σήμερα το πρωί, στι συνεδρία των συντονιστών, κάναμε μια συζήτηση για την ε, διαδικασία και όλες τις, ε, όλα τα θέματα της ε, συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην λήψη των αποφάσεων. Τώρα θα ακούσουμε τις διάφορες ομάδες που θα εκφράσουν τις απόψεις τους για τις προτάσεις που έχουν μπροστά μας και που έχουν προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις, μερικές φορές πολύ έντονες, ακόμα και στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Στις 2 Μαΐου θα ήθελα να πω ότι τα σχόλια ήταν μάλλον αρνητικά. Για να μην πω τίποτα πιο έντονο. Τώρα όμως μήπως θα πρέπει να πούμε και κάποια άλλα πράγματα και να μπούμε σε μια πιο επικριτική φάση ε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αυτά τα νούμερα ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά για την εκστρατεία, την προεκλογική για τις ευρωπαϊκές εκλογές του χρόνου. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε τώρα τους εισηγητές μας για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για τους ιδίους πόρους, άλλους εισηγητής για τους ιδίους πόρους, και ο Gerard Δεπρέ, ο οποίος είναι συνεισηγητής με τον κύριο Λεβαντόφσκι για τους ιδίους πόρους, μας εκπροσώπησαν την Δευτέρα το πρωί στις 14 Μαΐου, όταν έγινε η ενημέρωση της ομάδας γενικών υποθέσεων του Συμβουλίου. Και θα μας πει ποια ήταν η κατάσταση και τι κράτησε από αυτή την πρώτη ενημέρωση. Και συνεχεία θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές και σε όλους όσους θέλετε να πάρετε το λόγο για να μιλήσετε για αυτά τα θέματα. Ποιος θα μιλήσει, η Ιζαμπέλ Τωμά, ο κύριος Όλμπριχτ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όταν ήρθε εδώ ο Επίτροπο ε, την Κέρη, είπαμε και εμεί κάποιε παρατηρήσει, κάνουμε κάποιε παρατηρήσει, κάποια σχόλια. Ε, είπαμε τα προβλήματα που έχουμε. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί έκτοτε. Γιατί? Γιατί τα νούμερα τα οποία δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως η ανακοίνωση η οποία έγινε από την Κομισιόν για τα αριθμητικά στοιχεία του, επόμενου πουδουπού, όπως προετοιμάστηκε από την Κομισιόν, δεν μοιάζουν να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τι εννοώ. Τροποποιούμε κάθε φορά που θέλουμε να περάσουμε ένα νούμερο, κρύβουμε τον τύπο. Δηλαδή, Κάθε φορά που κάνουμε μία... Ε, θέλουμε να περάσουμε ένα νούμερο, μιλάμε για την Ευρώπη των 27 ή την Ευρώπη των 28. Ε, επίσης μιλάμε για κειμενόμενο, ευ, κειμενόμενα ευρώ ή μόνιμα ή σταθερά ευρώ. Ε, επίσης ε, βάζουμε το Ταμείο Ανάπτυξης ε, στο, στις οροφές ε, για να αλλάξουμε τα νούμερα του Πουδουπού. Μιλάμε για διάφορα κόλπα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερωτηματικό για την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα των ε, στοιχείων που μας δόθηκαν. Γιατί. Εδώ καταρχά θέλω να ευχαριστήσω τις ε, υπηρεσίες και του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν για τη δουλειά που κάνανε. Ε, γιατί πραγματικά φωτίζουν τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που ανακοίνωσε η Κομισιόν και σε αυτά που εμείς έχουμε μπροστά μας στο χαρτί. Φυσικά θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την Κομισιόν για να δούμε αυτά τα νούμερα και να μιλήσουμε για αυτά τα νούμερα. Φυσικά θα πρέπει να γίνει αυτό το περίφημο ραντεβού που έχουμε ζητήσει και που περιμένουμε απελπισμένα να μας ε, δοθεί από την Κομισιόν. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι να καταδεχτεί η Κομισιόν να έρθει εδώ και να μιλήσει ε, για τα νούμερα και να συγκρίνει τα δικά της με τα δικά μας. Θα βάζουμε στο κείμενο και κυρίως στο ψήφισμα των ομάδων που αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε στην επόμενη Ολομέλεια, θα βάλουμε τα νούμερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι να καταδεχτεί η Επιτροπή να μας πει κάτι και να κάνει τη σύγκριση. Είμαστε πιεσμένοι. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών με σοβαρότητα για το που δου που, χωρίς να έχουμε αυτά τα, σωστά, τα νούμερα, χωρίς να έχουμε τα σωστά νούμερα. Υπάρχουν και άλλα σημεία, πολύ σημεία. Δυστυχώς, με την πρόταση της Κομισιόν, ε, οι πολιτικές αλληλεγγύης διαλύονται, ε, έχει μείωση η πολιτική συνοχής. Βλέπουμε να ξαναγίνεται αυτό που έγινε στο τρέχον πουδουπού. Σε άλλους όμως προϋπολογισμούς. Ε, βγάζουμε από τη μία τσέπη και βάζουμε στην, ε, στην άλλη τσέπη. Ε, η μία τσέπη από την οποία βγάζουμε είναι η γεωργία κυρίως, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει φιλοδοξία, δεν υπάρχει σοβαρότητα, δεν υπάρχει σαφήνεια. Δεν υπάρχει θέληση στην πρόταση της Κομισιόν. Το είπα και χθε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Κοινωνικού Συμβουλίου η Κομισιόν ήξερε τι να περιμένει από το Συμβούλιο και τέθηκε κάπου στο, στο μέσο, ας πούμε, ανάμεσα στο Συμβούλιο και, στην, και στο Κοινοβούλιο. Ε, δεν, είχε φιλοδοξία, δεν είπε εγώ θέλω να υλοποιηθεί ένα project το οποίο είναι αυτό. Απλώς τέθηκε κάπου στη μέση έτσι. Διάλεξε να τοποθετηθεί στη χρυσή τομή ανάμεσα στο κοινοβούλιο και στο συμβούλιο. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρότασή της στο επίπεδο των φιλοδοξιών μας. Η κυρία Καλβινιού θα απογοητευτεί που δεν σας άκουσε κυρία Τωμά γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Νομίζω κατά τις 11 θα φτάσει. Αλλά μπορούμε να τις πούμε τι τις είπατε. Δεν υπάρχει σαφήνεια, δεν υπάρχει φιλοδοξία βασικά. Υπάρχουν, υπάρχει έλλειψη και στους δύο αυτούς τομείς. Ο κ. Όλμπριχτ έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα μόλις είπε η κυρία Τόμα. Παρατηρούμε και στο Συμβούλιο από τη μια μεριά την αντίθεση, την αντιπολίτευση, διότι είναι υπερβολικά μεγάλες οι περικοπές, από την άλλη μεριά πάλι αντίσταση, διότι λένε ότι οι περικοπές είναι πολύ περιορισμένες, πολύ μικρές. Είναι δύσκολο να λυθεί αυτό. Γι' αυτό η θέση μας θα πρέπει να εκφραστεί σήμερα και να είναι ότι θα απευθυνθούμε ως Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο δεν μπορούμε όμως να απευθύνουμε στο Συμβούλιο χωρίς να γνωρίζουμε τους ακριβείς αριθμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τώρα διαφορετικές αναλύσεις. Ποια είναι η πραγματική επίπτωση δηλαδή των προτάσεων της Κομισιόν. Και βέβαια να περιληφθεί σε αυτά και η ανάλυση του Κοινοβουλίου. Και τώρα βέβαια επιγόντως χρειαζόμαστε την ανάλυση ή τις αναλύσεις της Επιτροπής, της Κομισιόν. Γιατί, διότι εργαζόμεθα τώρα στο επίπεδο πολύ γενικών πληροφοριακών στοιχείων. Διότι η Κομισιόν, και αυτό για μας την Επιτροπή Προϋπολογισμών, είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε, ότι η Κομισιόν έχει αλλάξει την δομή του προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, ο ESF είναι ESF συν η e ΕΣΕΦ, σύν, όμως δεν είναι όπως ήταν πριν. Έχει πρόσθετα στοιχεία που δεν περιλαμβάνονταν στον ΕΣΕΦ e προηγουμένως. Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε τον σημερινό ΕΣΕΦ e με εκείνον που ήταν χθε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε επίσης την σημερινή συνοχή με την χθεσινή. Διότι και η συνοχή έχει αλλάξει. Το όλο κεφάλαιο της συνοχής έχει αλλάξει. Άρα υπάρχουν πολλά στοιχεία όπου χρειάζεται καλύτερη γνώση Invest EU. Τι σημαίνει συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα νούμερα και ποιο θα αναλάβει να το κάνει. Διότι έχουμε πληροφορίε ανατομέα, όπως και το πακέτο EMU και το πακέτο για την Ευρωζώνη. Όταν λέμε για δάνεια to -back και μέχρι 30 εκατομμύρια και ότι τα υπόλοιπα θα είναι από τις εθνικές συνεισφορές και διάφορα άλλα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Πρώτα θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για δομική αλλαγή, για αλλαγή φιλοσοφίας. Δεύτερο, ότι τα νούμερα χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο που να μην είναι σήμερα δυνατό να γίνει σύγκριση. Μπορούμε να προσπαθήσουμε εμείς οι ίδιοι. Αλλά για να το απλοποιήσω, όταν λέμε ότι έχουμε την πληροφορία μάλλον η συνοχή είναι, μάλλον η γεωργία είναι μείον 5, οι άμεσες πληρωμές μείον 4 και η συνοχή μείον 7. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να αρχίσουμε την ανάλυση και ιδίω όταν θα έχουμε την ανάλυση του Κοινοβουλίου που λέει ότι δεν είναι μείον 7, αλλά τουλάχιστον μείον 10. Και το Ταμείο Συνεχής μείον 45. Εάν το Ταμείο Συνεχής είναι μείον 45, αυτό σημαίνει ότι αυτό θίγει άμεσα τις χώρες συνοχής. Ίσως γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι χώρες συνοχής δεν θα είναι πλέον χώρες συνοχής. Αλλά εμείς δεν το γνωρίζουμε. Τέλο πάντων δεν είναι γνωστό αυτό. Ίσως ορισμένες να ξεπεράσουν το όριο του 90% του ΑΕΠ, του εθνικού επίπεδου. Αλλά ως, εφόσον, όσον δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα, είναι απλώς αριθμοί που χρησιμοποιούμε χωρίς να γνωρίζουμε τι κρύβεται από πίσω. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιγόντω συγκεκριμένες αναλύσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσει. και αμέσως μετά να αρχίσουμε να δουλεύουμε ε, στους, επί των τομέων και μετά αμέσως να συνεννοηθούμε με το Συμβούλιο. Συνεισηγητή τώρα των ίδιων πόρων, ο κύριος Λεβαντόσκη ή ο κύριος Δεπρέ. Λεβαντόσκη, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι συγκρίσιμα στοιχεία οφείλει να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σταθερές τιμές 2018. Δεν έχει γίνει αυτό ακόμη. Και όχι μόνο η πλευρά των δαπανών του προπολογισμού δεν είναι τόσο σαφής, δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά και η πλευρά των εσόδων. Γιατί έχουμε περίεργα νούμερα με ετήσιους μέσους όρους από το 2021 στο 2027 για να μπορούν να συζητηθούν αυτά τα πράγματα, για να μπορέσει να, συζητηθεί η πρόταση που κάνει η Κομισιόν για το ΠΔΠ, χρειαζόμαστε όντω συγκρίσιμα νούμερα, τα οποία δεν έχουμε. Εσείς κύριε Ντεπρέ. Κύριε Πρόεδρε. Προσθέτω δύο στοιχεία. Συμφωνώ με τον Λεβαντόφσκι για τους ιδίους πόρους και ανεξαρτήτως κάποιων πραγμάτων των οποίων η απουσία είναι ιδιαίτερα εντύπηρη. Δύο στοιχεία. Το γεγονός ότι εδώ και χρόνια ζητούμε μεταξύ των άλλων εσόδων που τροφοδοτούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης οι κυρώσεις που επιβάλλονται, πρόστιμα δηλαδή, στις επιχειρήσεις για μη σεβασμό τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ζητούμε εδώ και χρόνια να τροφοδοτούν τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντί να επιστρέφονται απλούστατα στι χώρε μέλη. Δεν εμφανίζονται όμω στι προτάσει τη Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να εξηγήσει, κομψιόν εννοώ πάντα, για ποιο λόγο δεν περιλαμβάνει αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο. Θα ήθελα να γνωρίζω επίσης γιατί ενώ το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει και με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της δυνατότητας επιβολής φόρου στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό τομέα, πάλι στις προτάσεις της Επιτροπής δεν περιλαμβάνεται. Και πιο, πιο ε, ε, συνολικά, ως και ο εισηγητής για, για τους ίδιους πόρους, έχω τρία στοιχεία. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες των άλλων συναδέλφων για τα νούμερα και για τη συγκρισιμότητα μεταξύ του μελλοντικού πλαισίου ΠΔΠ και του παρόντος. Όταν γίνονται αναλύσεις δεν μπορεί να έχει κανείς μια ξεκάθαρη ιδέα και γιατί, διότι δεν είναι πάντοτε οι ίδιες οι βάσεις για τη συγκρισιμότητα. Πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει να καταθέσει ένα έγγραφο τέλο πάντων το οποίο να επιτρέπει να κάνουμε πραγματικές συγκρίσεις. Δεύτερο, είναι σαφέ ότι θα υπάρχουν τρία κρίσιμα σημεία. Πρώτη, συνοχή. Δεύτερο, γεωρική πολιτική. Τρίτη, τρίτο, μηχανισμός αναστολής πληρωμών σε περίπτωση μη σεβασμού του κράτους δικαίου. Για την συνοχή νομίζω ότι οι περικοπές είναι πολύ σημαντικότερες από αυτές που περιλαμβάνονται στο έγγραφο. Άρα πρέπει να γίνει μια συζήτηση πραγματικά σοβαρή και σε βάθος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξαναλέω για να υπάρχουν, υπάρχουν δυνατότητες σύγκρισης. Για το κράτος δικαίου έχω μια έχω κάνει μια σκέψη. Έκανα μια σύντομη ανάλυση χωρίς να πω σε λεπτομέρειε του μηχανισμού με τον οποίο κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει να, και μάλιστα μέσα σε μια σταδιακή προσέγγιση, να διακοπούν τις πληρωμές. Σε ποια βάση θα γίνει αυτό, θα χρειαστεί όμως απόφαση του Συμβουλίου. Αλλά το Κοινοβούλιο δεν παίζει κανένα ρόλο. Είμαστε το ένα σκέλος της αρχής του προϋπολογισμού. Υπάρχει μια φράση γενικού χαρακτήρα που λέει «Α, ναι, το Κοινοβούλιο ε, ε, εμπλέκεται, ξέρω κάτι τέτοιο». Ε, δεν είναι πράγματα αυτά. Είμαστε το ένα σκέλος της αρχής του προπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει, βεβαίω, αλλά το Κοινοβούλιο δεν έχει απόλυτος τίποτα να πει. Πρέπει να κάνουμε πάλι μια σοβαρή συζήτηση για τον μηχανισμό αυτό. Θα περιοριστώ σε αυτά για την ώρα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις πλέον εισηγητές και πρώτος τον κύριο Φερνάντες. Θα μιλήσω πορτογαλικά κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου το λόγο. Δικαίως διευκρινίσαμε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και πραγματικά επισήλθαμε σε μεγάλο επίπεδο λεπτομέρεια. Νομίζω ότι εμεί θα πρέπει να δημοσιεύσουμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα, προκειμένου να εξηγήσουμε και τη μεθοδολογία που ακολουθούμε. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε περικοπή 40% στο Ταμείο Συνοχή. Αυτά τα ταμεία προορίζονται για τι πιο φτωχέ χώρε. Για όσου ε, έχουν ε, ανάπτυξη κατά κεφαλία ΕΠ κατώ από 90%. Η περικοπή των ταμείων συνοχής θα σημαίνει τέλος της συνοχής. Δεν θα υπάρχει λόγο να το αποκαλούμε ταμείο συνοχή πλέον, να το πούμε ταμείο κατά τη συνοχή. Δεν θα είχε οποιαδήποτε ε, χρήση, οποιαδήποτε ωφέλεια σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ε, διαφορών μεταξύ των περιφερειών. Περικοπή 25% για την ε, περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε περιφερειακή σύγκληση και συνοχή. Η ύπεθρος λοιπόν είναι σημαντική, σημαντικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Χωρίς αυτή δεν θα υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παρούσα μορφή της. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Ένωση θεωρώ ότι με την πρότασή της α, αντίκειται στην διακήρυξη Σούμαν χρειαζόμαστε συγκεκριμένε δράσει οι οποίες θα καταδείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Ο προπολογισμό 2001-2027 δεν είναι ένα προπολογισμό που θα δείχνει έμπρακτα αλληλεγγύη. Άλλο ένα θέμα, η διαφάνεια. Και εδώ περικοπές. 6,2, 7% και μετά μιλάμε για περικοπές πάνω από 10%. Όλα αυτά σε πολιτικές συνοχής. 20-25% στο Ταμείο Συνοχής, η Γεωργία πάνω από 15%, πάνω από 25% περικοπές σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να βελτιωθεί. Θα πρέπει να τροποποιηθεί μάλλον. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα μόλι δεσμεύτηκε ότι θα συμμετάσχει σε τεχνικέ συναντήσει για να εξηγήσει την ε, μεθοδολογία που ακολούθησε. Και στη συνέχεια φυσικά δεν ήρθε στι ε, συναντήσει αυτέ, δεν τήρησε τι υποσχέσει τη, όχι επειδή το Κοινοβούλιο δεν ήταν διαθέσιμο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Θα πρέπει να συγκρίνουμε αριθμητικά στοιχεία, σταθερές τιμές. Δεν μπορούμε να α, συγκρίνουμε αριθμητικά στοιχεία του 2011 με αριθμητικά στοιχεία του 2018 και σε αυτούς τομείς υπάρχουν σπάλματα. Δηλαδή, άμα πάρουμε ένα ευρώ από τη μία τσέπη και το βάλουμε στην άλλη, σημαίνει ότι έχουμε δύο ευρώ. άμα έχουμε ένα φάκελο με χρήματα, το να διάσουμε και θα βάλουμε σε άλλο φάκελο, το πρόβλημα είναι σαφέστερο. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαφάνεια, αλλά επίσης απαιτούμε να αποτυπώνουν στον προπολογισμό και οι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι να παραβιάζονται έτσι κατάφορα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε λέει ο κ. Βιώτη, είναι πολύ δύσκολη η συζήτηση. Πολύ περίπλοκη. Είναι περίπλοκη, γιατί όπως είπε και η κυρία Τομά, δεν έχουμε τα εργαλεία στα χέρια μας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πραγματικά. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές περικοπές στη συνοχή. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές περικοπές ε, στη γεωργική πολιτική. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν πραγματικοί Πραγματικέ και νέες επενδύσεις. Δεν υπάρχει σοβαρή απάντηση σε σχέση με τους ίδιου πόρους. Το Κοινοβούλιο έθεσε ερωτήματα για τους ιδίους πόρους, ε, αλλά δεν έλαβε απαντήσει, όπως είπε και ο κ. Ντεπρέ. Υπάρχει στο βάθος η εικόνα μία ευρωπαϊκή Επιτροπής και άρα μία ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει καμία φιλοδοξία για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Επομένως, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και περίπλοκα σήμερα. Το λέω για μας και για τα όργανα που εκπροσωπούμε. Η σημερινή ε, συνεδρίαση στην πραγματικότητα είναι μια άσκηση ρητορική δυνότητα παρά, μια πραγματική πολιτική συζήτηση. Γιατί το να συζητάμε μεταξύ μα έχει κανένα νόημα. Θα πρέπει να συζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπούμε στην ουσία των διαφόρων θεμάτων θα πρέπει να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες που υπάρχουν σε σχέση με τα νούμερα, όπως υπόθηκε. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που ακούσατε. Και αφού διασκεδαστούν οι ανησυχίες και αμφιβολίες για τα νούμερα, έχουμε το καθήκον να μπούμε στην ουσία πια, πέρα από τις ρητορίε. Ο κύριο Φερνάντες τα είπε όλα πολύ σωστά, όλα όσα αφορούν την πολιτική συνοχή. Τώρα θα ήθελα να προσθέσω ένα τελευταίο στοιχείο. Έχουμε το καθήκον να σεβαστούμε την αρχή της διαφάνειας. Διαφάνεια για τους πολίτες. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει δημόσια, θα πρέπει να γίνει μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση και να υπάρχουν και συγκρούσεις αν χρειαστεί. Αλλά θα πρέπει να, είναι, να γίνει μπροστά στα μάτια των πολιτών, όλων των ενδιαφερομένων πολιτών. Φαντάζομαι τώρα εδώ πάνε επιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Φαντάζομαι ότι όλοι σας, όπως και εγώ, είμαστε έμπλεοι ερωτήσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για αυτά τα, τα νούμερα. Γιατί νομίζω ότι βάζουμε ε, με αυτό το επόμενο πουδουπού την Ευρώπη σε μια φάση αβεβαιότητας. Εμείς θεωρούσαμε ότι πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ότι πρέπει να κάνουμε υπολογισμούς και να κάνουμε και κάποιες ε, μακροπρόθεσμες ας πούμε, προβλέψει, α πούμε. Τα κάνουμε αυτά εμεί, αλλά τα κάνουν και τα πανεπιστήμια, μικρομεσαίε επιχειρήσει κτλ. Δεν πρέπει να του αφήσουμε σε αβεβαιότητα. Γιατί αλλιώ πώ θα κάνουν επενδύσει. Επομένω, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει τα πραγματικά νούμερα, ούτω ώστε να μπούμε σε μια πολιτική συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση. γιατί μέθοδο μιλήσαμε αρκετά. Τώρα πρέπει να μπούμε στην ουσία. Σας ευχαριστώ. Και ο κύριος Κορβέλ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την αναγκαιότητα ε, επαρκών και αξιόπιστων αριθμητικών στοιχείων συζητήσαμε επαρκώ και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε άλλο. Δεν είναι δυνατόν να, ε, να κάνουμε μια σωστή συζήτηση επί σωστή βάση χωρί τα στοιχεία τέτοια. Και δεν χρειαζόμαστε μόνο αριθμητικά στοιχεία. Χρειαζόμαστε και τη βάση υπολογισμού των αριθμητικών στοιχείων αυτών. Γιατί όταν διαπιστώνουμε μεγάλε διαφορέ, ε, μπορεί να είναι καλά αιτιολογημένε αυτέ οι αλλαγέ. Αλλά αν δεν ξέρουμε του λόγου, πώ θα συζητήσουμε. Εικάζουμε απλά. Δεν είναι ο ρόλο μα να εικάζουμε. Κατά τα άλλα, πρέπει να ομολογήσω ότι όλα αυτά που άκουσα ε, θεωρώ ότι δεν εστιάζονται στην ουσία του θέματο. Όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρκετά φιλόδοξη Θεωρώ ότι το επιχείρημα αυτό δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθεται και κάνει κάποιους υπολογισμούς και λέει, κοιτάξτε, αυτά θεωρούμε ρεαλιστικά. Αυτά υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο, προφανώς. Μπορούμε να ζούμε σε μια φανταστική πραγματικότητα και να θεωρούμε ότι έχουμε πολλά χρήματα, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό θεωρώ ότι είναι απλά εσφαλμένο και θα ήταν λάθος ε, στη συζήτηση αυτή να λέμε «Α, να κάνουμε επενδύσεις προκειμένου να πάει καλά η οικονομία». Δεν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση. Η οικονομία τα πηγαίνει καλά. Μόνο εφόσον υπάρχουν ε, καλές ρυθμίσεις, όταν δίνεται στην οικονομία και στις επιχειρήσεις ε, σωστέ ευκαιρίε, προκειμένου να μπορούν να ανθίσουν. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε εμεί την οικονομία. Και νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε και λανθασμένες προσδοκίες στους πολίτες. Δεν μπορούμε να αναμειχθούμε λοιπόν εδώ. Ναι, βεβαίως και να επενδύσουμε σε τομείς όπου μπορούμε να έχουμε προστιθέμενη αξία. Στις υποδομές, στην έρευνα. Αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε ήδη σήμερα και να θέσουμε τις προτεραιότητές μας. Αυτό θεωρώ ότι είναι το έργο μας. Και θεωρώ ότι είναι λάθος να μην μιλάμε για χώρες που είναι καθαροί εισφορείς ή χώρες οι οποίες απλά λαμβάνουν μόνο χρήματα. Ε, δεν είναι ανταποκριτή στην πραγματικότητα γιατί υπάρχουν τέτοιες χώρες που εισφέρουν καθαρά. Και ενδεχομένως να μην υπάρχει η ομοφωνία γενικότερα για δαπάνη περισσότερων πόρων. Βέβαια, ούτε εμεί εδώ πέρα συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιε χώρε οι οποίε εισφέρουν και κάποιε οι οποίε ε, λαμβάνουν χρήματα, τα πράγματα είναι λίγο προκαθορισμένα και θα πρέπει να τα, πάρουμε, να τα λάβουμε υπόψη. Σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Ντεπρέ. Εν συντομία, πρόεδρε. Μια και ήδη έχω πάρει το λόγο Συμφωνώ με τους συναδέλφους που ζητούν συγκρίσουμε αριθμητικά στοιχεία για να μπορέσουμε να εργαστούμε επί σωστής βάσης. Και βλέπουμε, για παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε ό,τι αφορά την έρευνα έχουμε 13 με 15%, στο Rasmus Plus 17%. Μα θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η πραγματική βάση προκειμένου να προβούμε σε συγκρίσεις. Κατά δεύτερον, το είπατε και εσείς πριν από λίγο κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και ένα μεταμφιασμένο αν θέλετε σημείο εδώ στον προϋπολογισμό. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις οι αυξήσει δεν είναι αυξήσει, είναι αυξήσει ε, ψεύτικε. Γιατί πρόκειται για, στοιχεία, για δαπάνε που γίνονται στον αλλού στον προπολογισμό και τώρα απλά μεταφέρονται κατά τρίτον. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από τις ευρωεκλογέ. Αυτή είναι η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η επίσημη. Αλλά αν ε, κληθούμε να παρουσιαστούμε και να παρουσιάσουμε περικοπές ε, στο εκλογικό μας κοινό σε ορισμένε περιφέρειες τέτοιου τύπου όπως ε, αυτές που προτείνονται αυτή τη στιγμή, τι να σας πω. Καλή τύχη, σας εύχομαι. Ναι, λέει ο Πρόεδρος, είναι η αρχή της πραγματικότητας, θα έλεγα, όπως είπε και ο κ. Κορμπέλ, του ρεαλισμού. Ο κύριος Σολέ. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε, είναι δύσκολο να τοποθετηθούμε με σαφήνεια έναντι της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν έχουμε βασικές δυσκολίες για τη σύγκριση των αριθμητικών στοιχείων. Όταν δεν έχουμε τα πλήρη στοιχεία και δεν γνωρίζουμε τα προβλήματα επακριβώς. Τούτου λεχθέντους. Υπάρχουν και κάποια ενδιαφέροντα σημεία στην πρόταση. Αλλά συνολικά θεωρούμε ότι είναι μια ευκαιρία η οποία χάθηκε. Την έχασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανησυχούμε. Αξιολογούμε διαφορετικά βεβαίως τα διάφορα σημεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά η βασική μας ανησυχία εστιάζεται στο εξή. Μάλλον σε τρία στιγμία. Καταρχάς, στον όγκο. Είμαστε βέβαιοι ότι ο παρόν προπολογισμό δεν επιδεικνύει επαρκέ επίπεδο φιλοδοξία και η συνολική αύξηση τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 0,8%. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένη αυτή η αύξηση δεδομένων φυσικά και των προκλήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και των πολιτικών φιλοδοξιών που έχουμε θέσει ή που πρέπει να θέσουμε. Άρα, ο Όγκος τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής απέχει παρασάγκα από αυτά που προτείνουμε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο 1,3% ήταν η δική μας πρόταση. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη, Νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο να τονίσουμε την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική συνοχή θα περιοριστεί, θα περικοπεί. 5% και το ESF Plus, το κοινωνικό ταμείο, εντάξει δεν λέω, σημειώνει μια μικρή αύξηση. Ανεπαρκέστατη όμως δεδομένου του ότι εξαφανίζεται ουσιαστικά η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και ουσιαστικά ενσωματώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο ESF. Είναι πραγματικά πολύ αδύναμη η προσέγγιση πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ε, ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτος τομέας ανησυχίας για την ομάδα μας η στρατιωτικοποίηση του προπολογισμού 17 δις ευρώ σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τροπής, τα οποία θα δαπανηθούν στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Τώρα για το τι με Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπιζόμαστε την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας, τις οποίες και εγκρίναμε πριν από κάποιους μήνες. Θα πρέπει να προσπιστούμε τα βασικά μηνύματα των προτάσεων αυτών και για μένα αυτό που είναι πολύ σημαντικό, γιατί άκουσα και τις συζητήσεις στο Συμβούλιο, θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε στεναρά τις δύο προτάσεις αυτές, όπως τις υποστηρίζαμε και πριν από κάποιους μήνες που τις εγκρίναμε στην Ολομέλημα. Για να δείξουμε ότι θα υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια έναν πιο δυναμικό προπολογισμό. Ευχαριστώ κύριε Σαντή. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα τους συναδέλφους που θεωρούσαν ότι αυτή η συζήτηση δεν έχει νόημα. Γιατί δεν έχουμε τα πραγματικά νούμερα. Εγώ δεν συμφωνώ 100%. Υπό την έννοια ότι οι κατευθυντηρίες γραμμές για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο κατά την Κομισιόν είναι ξεκάθαρες. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε τα πραγματικά νούμερα για να αποφανθούμε οριστικά. Αλλά οι κατευθυντήριε γραμμές νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρες και αρκετά δηλωτικές. Και εγώ ακριβώς γι' αυτό είμαι ανήσυχο και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η πρόταση. Και είναι πολύ διαφορετική και πόρα απέχει από αυτό που θα ήθελαν οι πολίτες. Και κάποιο είπε προηγουμένω ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο, μέσα στο 2019, με αυτή την πρόταση, πώ θα πάμε σε ευρωεκλογέ. Πρέπει να κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια, ούτω ώστε αυτό το επόμενο πουδουπού να έρθει πιο κοντά σε αυτό που επιθυμούν οι πολίτε. Τώρα, κάποια πιο συγκεκριμένα σχόλια. Το πρώτο που δεν έχει νόημα κατά την απόψή μου είναι το να δούμε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο αυξάνεται το οποίο ε, τη στιγμή που οι πολίτες ξέρουν ότι από το Μάρτιο του 2019 τα κράτη-μέλη από 28 θα γίνουν 27. Μερικές φορές γίνεται λόγος για διαχείριση του προϋπολογισμού των κοινωτικών οργάνων με τον ίδιο τρόπο που ένας πατέρας, ας πούμε, διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα πατέρα που βλέπει ότι η οικογένειά του από πέντε σε τεσ... Ε, που γίνεται από πέντε μέλη τέσσερα, στην πραγματικότητα ξέρει ότι έχει λιγότερου πόρου στα χέρια του για να ξοδέψει εν συνεχεία. Αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη μα, δεν το καταλαβαίνω λοιπόν. Εγώ θα περίμενα έναν προπολογισμό μειωμένο ε, σε νούμερα. Τώρα για τι κατευθυντήριε γραμμέ που προτείνει η Κομισιόν. πολιτικό πώ. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο το γεγονό ότι ορισμένα ταμεία ουσιαστικά αποφασίζεται η μοίρα τους με βάση τις πολιτικές σκέψεις και συμφέροντα κάποιων κρατών μελών. Ο Γιούγκερ και ο Ότιγκερ ε, στην Ολομέλεια μας εγγυήθηκαν ότι η ιστορία του του κριτηρίου του κράτους δικαίου δεν εφευρέθηκε για να τιμωρήσουμε κάποια κράτη-μέλη. Ξέρουμε ποιε είναι οι διαδικασίε σήμερα και ποιες ε, διαδικασίες τρέχουν ήδη εναντίον δύο κρατών μελών. Μας ανησυχεί αυτό το θέμα. Επίσης, με ανησυχεί το θέμα των ταμείων σταθεροποίησης για την Ευρωζώνη και τι μεταρρυθμίσει. Το να υποχρεώσουμε κάποια κράτη-μέλη, να πούμε σε κάποια κράτη-μέλη, σου δίνω κάποια λεφτά εάν κάνεις τις μεταρρυθμίσεις που θέλω εγώ, μου φαίνεται εκβιασμός. Είναι μια μορφή εκβιασμού που δεν νομίζω ότι προσάδει σε αυτά τα θεσμικά όργανα. Ακόμα και για την ΚΑΠ και για την ε, συνοχή θεωρώ ότι η πρόταση είναι απαράδεκτη. Περιμένω τα πραγματικά νούμερα. Αλλά νομίζω το να ε, δυσκολέψουμε έτσι περαιτέρω την κατάσταση της γεωργίας που ήδη είναι σε δύσκολη κατάσταση γιατί ας πούμε βλέπω στην Ιταλία τι γίνεται. Επηρεάστηκε πάρα πολύ η Ιταλική γεωργία από, τις, ε, από τα αντίμετρα της Ρωσίας. Εάν μειώσουμε ακόμα τον προπολογισμό της ΚΑΠ θα ήταν καταστροφικό για την Ιταλία. Ε, στην Ιταλία η γεωργία μετράει πάρα πολύ στο ΑΕΠ. Σε άλλα κράτη-μέλη, ειδικά στα πιο ανεπτυγμένα ας πούμε, η γεωργία βαραίνει λιγότερο, αλλά βαραίνει ακόμα αρκετά σημαντικά στο ΑΕΠ. Επομένω, νομίζω ότι θα μπορούσαν θα μπορούσαν αυτέ οι περικοπέ να είναι αποσταθεροποιητικέ για διάφορε οικονομίε. Για την πολιτική συνοχή, το ίδιο. Δεν θα επηρεαστούν μόνο οι χώρε οι οποίε έτσι είναι ανάπτυξη, ας πούμε, ή τις περιφέρειες που είναι υπό ανάπτυξη, αλλά θα επηρέαζει ακόμα και περιοχές που σήμερα χρησιμοποιούν αυτά τα ταμεία για να αυξήσουν έτσι περαιτέρω την ανάπτυξή τους. Τώρα, για την άμυνα. Το να έχουμε ένα τέτοιο προπολογισμό, όταν βλέπουμε ότι τα διεθνή στοιχεία μας βλέπουν ότι οι απόψει των κρατών μελών για τα καυτά θέματα της εξωτερικής πολιτικής είναι διαφορετικές, ε, είναι προβληματικό. Επίσης, τα διοικητικά έξοδα, δεν το καταλαβαίνω καθόλου αυτό το σημείο. Από τις πρώτες ε, συζητήσεις και από την πρώτη πρόταση, βλέπω ότι τα διοικητικά έξοδα μέσα σε αυτή την εφταετία θα είναι σημαντικό κομμάτι. Δεν μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες να καταλάβουν γιατί τόσα πολλά έξοδα. Επίσης, για τα κονδύλια, τα προενταξιακά. Και εδώ υπάρχει δυνατότητα αύξηση. Ιστορικά αυτά τα ταμεία, ξέρετε πολύ καλά ότι το 40 με 50% τους πήγαινε στην Τουρκία δεδομές της ε, διεθνούς κατάσταση, ακόμα και του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε με την Τουρκία, εγώ θα έκανα μια διαφορετική ας ανάλυση για αυτά τα ποσά που πηγαίνουν στην Τουρκία. Γιατί μου φαίνεται ότι είναι... δεν είναι σωστό να τιμωρήσουμε διάφορους ή να χρησιμοποιήσουμε το, το κριτήριο του κράτους δικαίου ας πούμε, για να τιμωρήσουμε δικά μας κράτη-μέλη και να δίνουμε τα ίδια ποσά ας πούμε, στην Τουρκία η οποία προφανώς δεν σέβεται το κράτος δικαίου. Πολύ ωραία, τελειώσαμε τους κοιόδους εισηγητές. Euh, Και τώρα λοιπόν να, να επιβεβαιώσουμε τις αποφάσεις που λάβαμε σε ό,τι αφορά τους συντονιστές. Να αποστελούμε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Επιτροπό, γιατί ο Επιτροπός ε, όταν ε, ήλθε στην Επιτροπή μας στις 3 Μαΐου είχε δεχτεί να γίνει συνάντηση των ομάδων μα από την επόμενη Δευτέρα για να υπάρξει μια συγκρισιμότητα σαφής των ε, αριθμητικών στοιχείων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Σημειώθηκε καθυστέρηση και στην καθυστέρηση αυτή λοιπόν διαμαρτυρόμεθα με την επιστολή την οποία θα αποστείλω προς τον Επιτροπό Έττιγκερ σήμερα το απόγευμα. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στην ε, διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Υποστηρίζω την προσέγγιση των συναδέλφων που μίλησαν πριν, ότι δηλαδή χρειαζόμαστε αναγκαία συγκρισιμότητα. Προτείνω, εάν είναι δύσκολο να γίνει αυτό στο τεχνικό επίπεδο, να επαναλάβουμε, μια διαδικασία που είχαμε εκτελέσει στην αρχή της θητείας. Δηλαδή, να οργανώσουμε ένα σεμινάριο με συμμετοχή βουλευτών, διότι θεωρώ ότι θα μας δώσει την ευκαιρία να θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα τεχνικού χαρακτήρα και θα έχει ενδιαφέρον να ζητήσουμε να έρθει και το τμήμα, το ευρωπαϊκό τμήμα του Συμβουλίου. Όταν δηλαδή μιλούμε για ζητήματα συγκρισιμότητας, είναι κρίσιμο να έχουν μια ερμηνευτική βάση συγκρισιμότητας και τα τρία θεσμικά όργανα. Δεν θέλω να φτάσουμε να καθίσουμε σε τριμερή διάλογο και να μιλούμε και να μαλώνουμε επί ώρες με τους εκπροσώπους των δύο άλλων θεσμικών οργάνων για το ποια νούμερα είναι συγκρίσιμα και ποια όχι. Και σημειώνω ότι αυτό το έχουμε ζήσει ήδη ορισμένες φορές. Είναι ένα θέμα αυτό. Τονίζω εξάλλου ότι δεν είναι αναγκαία ότι τα κίνητρα είναι όλα η στεροβουλία από πλευρά των άλλων θεσμικών οργάνων. Βεβαίω και παίζει ένα ρόλο η Βρετανική αποχώρηση. Σε ένα σεμινάριο που συμμετείχα τελευταία και ήταν παρούσα εκπρόσωπος της Λιθουανικής Πρεσβείας, η οποία ανακοίνωσε ότι η χώρα τη, η Λιθουανία, πάει να γίνει σιγά σιγά καθαρο συνεισφορέα και βεβαίως μπορώ να το φανταστώ ότι αυτό είναι αλήθεια. Διότι μειώνεται ο μέσος όρος του καθαρού εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν αποχωρήσει μια χώρα όπως η Μεγάλη Βρετανία. Θα είναι πολύ χαμηλότερη λοιπόν η τιμή από αυτή που γνωρίζουμε από το μέχρι τώρα πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Και βεβαίως και οι ροές θα είναι διαφορετικές. Γι' αυτό προσοχή. Εάν οργανώσουμε αυτό το σεμινάριο για τη συγκρισιμότητα θα είναι σαν να τραβήξουμε στην άκρη μια κουρτίνα και να δούμε πραγματικά ποια είναι η εικόνα, η πραγματικότητα. Πρέπει να δούμε λοιπόν. Ναι μεν έχουμε την επιθυμία ε, να έχουμε συγκρίσιμα νούμερα. Σύμφωνα απόλυτα. Υπάρχουν όμως βάσεις υπολογισμών που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μετακινούνται, δεν είναι απόλυτα σταθερές. Και το Υπουργείο Οικονομικών στο Βερολίνο έχει κατατρομάξει την κοινή γνώμη σχετικά με το πόσο θα αυξηθεί η γερμανική συνεισφορά. Και μάλιστα περιλαμβάνονται και στη συμφωνία που έχουν κάνει τα κόμματα του μεγάλου συνασπισμού. Σε αυτά συμμετείχα και εγώ όταν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για την δημιουργία του Εβραίου Συνασπισμού είναι και σοσιαλδημοκράτης ο Υπουργό Οικονομικών στο Βερολίνο, που ακολουθεί στα χνάρια του Σόιπλε και κάνει ό,τι έκανε και αυτός. Και βάζουν μέσα στα 7 χρόνια και τον πληθωρισμό και λένε ότι αυξήθηκε η συνεισφορά της Γερμανίας κατά 28% χωρίς να είναι αναγκαίο ότι ε, συνέβη αυτό. Γνωρίζουμε ε, αυτά τα πράγματα. Τώρα, με ναι μεν έχουμε την επιθυμία για συγκρισιμότητα, αλλά μην λησμονούμε και αυτά που σας εξήγησα. Και είναι σημαντικό ε, να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές χρηματοοικονομικές ροές και ορισμένοι είπαν ότι κάποια πράγματα δεν τους αρέσουν, αλλά πρέπει να δούμε ποιο είναι το τροποποιημένο περιεχόμενο των προγραμμάτων και γι' αυτά δεν άκουσα ακόμα τίποτα. Τώρα, μία ακόμα παρατήρηση για καθαρούς εισφορείς και καθαρούς δικαιούχους, χώρες δηλαδή. Αυτή η συζήτηση είναι παροχημένη, είναι του 20ου αιώνα. Βεβαίω υπάρχουν, βλέπω ο κύριος Κιόλμελ αποχωρεί, υπάρχουν χρηματοπιστωτικές ροές που δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν. Το αεροδρόμιο των Αθηνών που χτίστηκε για να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγινε από μια, χτίστηκε δηλαδή από φύρμα τη εκλογική μου περιφέρεια, της ΕΣΥΣ, με χρήματα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό λοιπόν πήγανε στον ελληνικό προπολογισμό και από τον ελληνικό προπολογισμό στι τσέπε τη Χόχτιφ, με, η οποία λειτουργήσε βεβαίω και με θηγατρικέ. Οι χρηματοπιστωτικέ αυτέ ροέ δεν είναι πλέον μετρήσιμε. Δείχνουν όμω ότι υπάρχει όντω ένα ενιαίο οικονομικό χώρο, όπου η συζήτηση για το ποιο πληρώνει και ποιο παίρνει, από ποια τσέπη βγαίνουν και ποια τσέπη μπαίνουν, τελικώ είναι η συζήτηση αυτή παροχημένη. Και σιγά σιγά είναι αναγκαίο να το αντιληφθούμε αυτό και να αντιληφθούμε ποια είναι η πραγματικότητα μια κοινή αγορά. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Η κυρία Καλβίνιο έχει έλθει στο μεταξύ και ρωτώ αν επιθυμεί να λάβει το λόγο τώρα. Μ' όμω δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω την κυρία Τωμά όταν τοποθετήθηκε λίγα λεπτά πριν να έρθετε. Μήπω η κυρία Τωμά μπορεί μέσα σε μισό λεπτό. Ε, ποια ήταν η πραγματική πεμπτουσία των λόγων της. Νόμιζα θα το κάνετε εσείς κύριε Πρόεδρε. Αλλά ευχαρίστως. Το πρόβλημα κύριε Καλβίνιο, το οποίο αντιμετωπίζουμε, είναι ότι έχουμε την εντύπωση ότι μεταξύ των λόγων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αριθμών που προβάλλει υπάρχει μια μικρή αλλά ίσως και μια μεγάλη απόσταση. Υπάρχει ένα πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, διότι τα νούμερα από τη στιγμή που τα βάζουμε κάτω και τα εξετάζουμε, δεν μας φαίνονται πάντοτε αξιόπιστα. Ενώ δηλαδή ότι πρώτα έχουμε χρήση ε, κειμενόμενου ευρώ ή τρέχοντος ευρώ και όχι σταθερού ευρώ, ε, σε αυτό ίσως ε, δεν, θα, θα, λάβουμε ως βάση τα νούμερα της Ευρώπης των 27 ή των 28 ε, αυτό μπορεί να συμβαίνει για τον τομέα της για άλλα και για την οροφή που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Α114 για την επανένταξη τώρα για το 108 για το μελλοντικό ε, δημοσιονομικό πλαίσιο αυτά δεν είναι σαφή αυτό που θα θέλαμε, εν πάση περιπτώσει, κυρία Καλβίνιο, και το έχουμε ήδη πει και στον Επίτροπο κ. Έτιγκερ, θα θέλαμε δηλαδή να διεξαχθεί μια σοβαρή συζήτηση επί της μεθοδολογίας, επί των αριθμητικών στοιχείων, επί του συνόλου δηλαδή των αριθμητικών στοιχείων που μας έχουν υποβληθεί, να μπορέσουμε να συζητήσουμε σοβαρά, για να έχουμε μια όσο το δυνατόν ε, πιο αντικειμενική ενατένιση ε, Τη πραγματικότητα, διότι τα όσα ε, έχουμε... Α, αυτά που είπατε προηγουμένως ήταν κάπως πιο αυστηρά, πιο αγριοπά. Χάσατε την ε, πρώτη εκδοχή, κυρία Καλβίνιο. Ορίστε, κυρία Γενική Διευθύντρια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μην ανησυχείτε, ήδη με είχαν ενημερώσει η συναδελφοί μου για τον τόνο και το ύφο τη πρώτη παρεμβάσεω. Πάντω, ευχαριστώ πολύ την κυρία Τομά η οποία ε, φέρεται πάντοτε με ιδιαίτερη ε, ευγένεια και αξιοπρέπεια. Βεβαίω όλοι βρισκόμαστε... Α, θα συνεχίσω όμω στα αγγλικά. Είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων στον κύριο Γκάιερ και λυπούμε που αποχώρησε, διότι νομίζω ότι έφεσε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Δηλαδή, συζήτηση περί διαφάνειας, συγκρισιμότητα κλπ. Και επιτρέψτε μου να πω τρία πράγματα τώρα για να απαντήσω στα σχόλιά σα. Πρώτα, Κοιτάξτε, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες αριθμών και κάνουμε, ή μπορούμε να κάνουμε υπολογισμού με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Και πιθανώ όλοι οι υπολογισμοί αυτοί που θα κάνουμε να είναι και σωστοί. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε το έργο, το δικό μα και το δικό σα όντας όσο γίνεται πιο διαφανής στις προτάσεις της Κομισιόν. Συμφωνώ όμως ότι θα χρειαστεί και άλλη τεχνική εργασία. Κατανοώ ότι οι τεχνικές συζητήσεις προβλέπονται ήδη για τις 24 Πέμπτου, όπου θα διεξαχθεί η τεχνική συζήτηση. Ευχαρίστως όμως να έλθω και να σας κάνω μια παρουσίαση, όπως θέλετε εσείς, όπως αποφασίσετε. Ε, έχουμε τη διάθεση δηλαδή και είμαστε και έτοιμες να ε, δείξουμε απόλυτη διαφάνεια απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βεβαίω όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στο Συμβούλιο υποβάλλονται εκ παραλλήλου και στο Κοινοβούλιο. Σε ό,τι μα αφορά λοιπόν, πλήρη σαφήνεια και απόλυτη ισότιμη μεταχείριση των δύο εταίρων θεσμικών οργάνων Συμβουλίου Κοινοβουλίου. Εργαζόμαστε τώρα επί του πίνακα συγκρισιμότητα. Όπω είπε όμω ο Γιάννη θα πρέπει να είμαστε προσεκτικέ, διότι περνούμε από έναν προπολογισμό τη Ευρώπη των 28 σε προπολογισμό τη Ευρώπη των 27. Και ειλικρινώ είναι ένα άλλο κόσμο. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα το οποίο προσπαθεί να περάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα σύγχρονο προπολογισμό μια μελλοντική Ευρώπη των 27. Δεν ήταν σωστό λοιπόν να πάρουμε τα νούμερα σαν δίθεν να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Και εκτός αυτού έχουμε απροποιήσει σημαντικά τον προπολογισμό και έχουμε απροποιήσει και τα προγράμματα. Άρα ορισμένα προγράμματα δεν είναι τα ίδια ε, όπως στο τρέχον πι όχι όμως για να προκαλέσουμε καμιά σύγχυση, αλλά για να τα αποκριθούμε στα όσα ζητείτε και εσείς, δηλαδή ένα πιο εύληπτο, πιο ευανάγνωστο προπολογισμό και πιο ευθυγραμμισμένο με τις πολιτικές προτεραιότητες. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το επιτύχουμε αυτό. Ξαναλέω, ευχαρίστω να έλθω να σας εξηγήσω ποιε αλλαγέ έχουμε κάνει στην αρχιτεκτονική του προπολογισμού. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε σε ό,τι αφορά συνοχή και γεωργία, που αντιλαμβάνομαι ότι είναι οι τομείς που σας απασχολούν περισσότερο, είναι πιο ευαίσθητοι και ο κύριος Ντεπρέ το ξεκαθάρισε αυτό απολύτως, βεβαίω δεν έχουμε καμιά ασφαλμένη δίποση σχετικά, είναι να πάρουμε το τρέχον δελταπί, να πάρουμε το έτος 2020, που είναι και το υψηλότερο του τρέχοντος πιδελταπή, σε τρέχουσες τιμές, και να αφαιρέσουμε την συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Για ορισμένα προγράμματα αυτό είναι κάπως πιο εύκολο. Εκεί όπου υπάρχει εθνική κατανομή, όπως γίνεται με τη, τα πράγματα της Γεωργίας. Αλλού χρησιμοποιούμε εκτιμήσεις. Πρόκειται για εκτιμήσεις. Γι' αυτά δεν τα έχουμε βάλει και σε ε, επίσημα έγγραφα. Πρόκειται για υποθέσεις. Και στη βάση αυτή έχουμε υπολογίσει τις αλλαγές. Και αυτά είναι τα νούμερα τα οποία κοινοποιήσαμε ή τέλο πάντων ανακοινώσαμε δημοσίω. Θέλω να τονίσω ότι δεν θα πρέπει να αντιδράσουμε υπερβολικά χωρίς να λάβουμε υπόψη το πολύ αυτό σημαντικό στοιχείο ότι δηλαδή θα πρέπει να βγει εκτός παρελθέσεως το Ηνωμένο Βασίλειο για το επόμενο ΠΔΠ. Δεύτερο σχόλιο. Α μην ρίχνουμε όλο το βάρο αν και αντιλαμβάνομαι την ελκυστικότητα του ποσοστού ΑΕΠ. Αυτό που λέμε στις χώρες μέλη είναι όμως και όλες οι χώρες μέλη άλλωστε εκπροσωπούνται και εδώ παροιμήν να μην χρησιμοποιούν αυτό το, το, το τεμ του 1% το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες αλλά και διότι το ΑΕΠ αλλάζει. Γιατί δεν και καλά να κρατάμε οπωσδήποτε ένα ποσοστό. Για να είμαι ειλικρινής, τα ποσά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφέροντας το 1,14% του ΑΕΠ στην βάση των υπολογισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν την επόμενη μέρα από την υποβολή της προτάσεως. Αν έχουμε τα ίδια νούμερα σε σύγκριση με τις προβλέψεις του προηγούμενου φθινοπόρου, ίσως θα ήταν 1,15 ή 1,16. Παρακαλώ λοιπόν να μην κολλάμε στο 1,13 ή στο 1,3 μάλλον. Και τι γίνεται αν η πρόβλεψη μειωθεί για το μέλλον. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταθέσουμε μια πρόταση, την οποία εμείς ε, παρουσιάζουμε ως ρεαλιστική. Αύξηση σε ονομαστική αξία κατά 15%. Το οποίο τα πει συν το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο είναι αύξηση περίπου 15% σε τρέχουσε τιμέ και ανταποκρίνεται λίγο πολύ στον προβλεπόμενο πληθωρισμό. Πρόκειται δηλαδή για ένα πληθωρισμό ο οποίο διατηρείται σταθερό. Σε σταθερέ τιμέ είναι ισοδύναμο. Ξεκινούμε όμω από μια Ευρώπη των 28 για να πάμε σε Ευρώπη των 27. Και ο προπολογισμό ω Τέτοιο διατηρείται σε σταθερέ τιμέ στο ίδιο επίπεδο. Μπορεί να το δει λοιπόν κανεί από διαφορετικέ πρόπτικε. Μπορεί να πει κανεί ότι είναι ρεαλιστικό, μπορεί να πει κάποιο να πει ότι είναι και φιλόδοξο. Γιατί περνάμε από Ευρώπη 28 σε Ευρώπη 27 με τον ίδιο προπολογισμό, Χωρί το κατεβάζουμε. Και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων κάποιε χώρε μέλη, πολλέ χώρε μέλη είπαν μικρότερη ένωση, μικρότερο προπολογισμό. Αυτό όμω δεν ανταποκρίνει στην πρόταση Κομισιόν. Ήθελα λοιπόν να σα δώσω κάποια σημεία αναφορά στη συζήτηση. Το τρίτο σχόλιο έχει ως εξής. Καταβάλαμε σημαντική προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε δικαιοσύνη και ισορροπία. Είναι σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό και για το όσο συζητούμε με τις 27 χώρες μέλη. Ο Επίτροπος τόνισε κατά επανάληψη ότι το κενό του Brexit που θα έχουμε στο πλευρά των εσόδων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 100% μείωση του προπολογισμού. Αυτά τα είπα και προηγουμένω. Παίρνουμε λοιπόν αυτή την προσέγγιση 50-50. Μισό από το κενό γίνεται περικοπή και μισό από το κενό είναι νέο χρήμα. Αυτή είναι η προσέγγιση στην οποία βασίζεται η πρόταση της Κομισιόν. Και μαζί με αυτό είπαμε, πρόκειται για μια έντιμη πρόταση και χωρί βάση για επιστροφέ. Και εμεί προτείνουμε να αφαιρεθούν οι επιστροφέ. Κάτι που είναι επίση σωστό, όπω είπε ο Γιάννη Κάιερ, είναι ότι ο υψηλότερο αυτό προπολογισμό σε ονομαστικέ τιμέ, σημαίνει και αύξηση των εθνικών συνεισφορών για τον πρώτο χρόνο. Ε, γι' αυτό προτείνουμε και αυτό ο μηχανισμό σταδιακής κατάργηση. Δεν είναι όμω ζήτημα μόνο εντιμότητα, είναι για να αποφύγουμε το άλμα από τη μια χρονιά στην άλλη. Για εμά, εν πάση περιπτώσει, και μαζί με την πρόταση για νέους ιδίους πόρους που γνωρίζω πόσο πολύ σας ενδιαφέρει και έχει κάνει σημαντική προσπάθεια να κάνει σχετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μας πάντως εντιμότητα και ισορροπία, η δικαιοσύνη και η ισορροπία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Και όταν συζητούμε κάποιε από τις χώρες μέλη του λέμε ότι όταν εξετάζουν την αύξηση των εθνικών συνεισφορών, δεν θα πρέπει να τις λαμβάνουν με ονομαστικές τιμές. Να πούνε, κοιτάξτε, ναι, είπε προηγουμένως για 30% δεν είναι σωστό να εξεταστεί με τον τρόπο αυτό, διότι πρόκειται για ένα προπολογισμό επταετία και σε αυτά τα 7 χρόνια θα υπάρξει και πληθωρισμό, θα υπάρξει και αύξηση του ΑΕΠ. Υπάρχει και ένα στοιχείο από την κατάργηση των επιστροφών και την επανεξισορρόπηση των εσόδων από τον Brexit και πρόσθετο εισόδημα. Αλλά μην τα ανακατεύετε όλα αυτά μαζί. Του λέμε λοιπόν, δέστε τα σε πραγματικού όρου. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι μιλώντα με πραγματικού όρου και με ονομαστικού όρου, είναι σωστό. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι να εξετάζει κανεί την ίδια πραγματικότητα. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή τη βάζει ονομαστικού όρου και καταθέτουμε του πίνακε και σε ονομαστικού και σε πραγματικού όρου. Μου λέτε, θέλουμε τα σημεία αναφορά. Αυτά επεξεργαζόμαστε τώρα. Ποιε θα είναι οι καλύτερε εκτιμήσει που μπορούμε να δώσουμε στις δύο, στα δύο σκέλη της αρχής του προϋπολογισμού για να κάνουν τους υπολογισμούς τους. Αλλά πρόκειται για νέο προϋπολογισμό, για μια νέα διαφορετική Ευρώπη, Ευρώπη των 27 και με διαφορετική αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η σύγκριση λοιπόν ή τέλος πάντων η απόλυτη στόχευση μόνο στη συγκρισιμότητα είναι κάπως παραπλανητική. Θα δώσουμε όμως εμείς, θα προσφέρουμε πλήρη διαφάνεια και όπως είπα και στην αρχή Είμαι απολύτως διατεθειμένη να έλθω να σας κάνω μια παρουσίαση, να σας δώσω και κάποια στοιχεία, τα οποία ίσως να μην είναι ορατά όταν εξετάζετε και όταν μόνο τους πίνακες και την ανακοίνωση, αλλά πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί εμείς συντάσσουμε τώρα και την νομική βάση για τις επόμενες εβδομάδες. Τούτε εδώ, τούτες εδώ μέρες το κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Γενική Διευθυντή. Η μικρή μας απογοήτευση οφείλεται στο γεγονός ότι όταν ο Επίτροπος ήρθε να παρουσιάσει το προϋπολογισμό 5η 3 Μαΐου, είχε δεσμευτεί ότι η ομάδα σας και η δική μας ομάδα της Γραμματείας της Επιτροπής Προϋπολογισμών θα μπορούσαν να συναντηθούν την επόμενη Δευτέρα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουν το κατά πόσο υπάρχει σύγκριση των ε, δικών μας και των δικών σας νούμερων. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Δεν συναντήθηκαν οι δύο ομάδες. Αυτό μας απογοήτευσε. Εξού λοιπόν και αυτή η συζήτηση που είναι έμπλεη αμφισβητήσεων, υποψία κτλ. Πότε πιστεύετε θα μας δοθούν κάποια αδιαμφισβήτητα νούμερα και που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε μια πραγματική σύγκριση για να αρθούν όλα τα ερωτηματικά και οι αμφιβολίες. Όταν υπολογίζετε το ποσό για την πρόοδο των ε, πιστώσεων του ορίζοντα 2020, αφαιρείται τα, τις πιστώσεις που κάθε χρόνο πήγαιναν προς τα βρετανικά εργαστήρια. Είναι σωστή αυτή η προσέγγιση, δεν είμαι σίγουρη, σίγουρος. Φυσικά, ε, έτσι μας δείχνετε ότι υπάρχει μια πρόοδος, αλλά ξεχνάτε τους διαγωνισμούς που είχαν ξεκινήσει. Και ξέρετε ότι τα βρετανικά εργαστήρια πολύ συχνά ήταν τα καλύτερα Επομένω, έχουμε κάποιε βάσει σύγκριση, κάποια νούμερα τα οποία μπορεί να τα αμφισβητήσει κανεί. Πολύ ωραία. Επανερχόμαστε στα ερωτήματά μα και θα δώσω το λόγο στην πρόεδρο Γκρέσλε. Πρόεδρε, θα ήθελα για να επανέλθω στη συζήτηση των συναδέλφων να διευκρινίσω το εξή, ότι η επιθυμία για πιο πολλά χρήματα είναι κατανοητή. Αλλά το θέμα είναι πού θα τη θέσουμε τα χρήματα αυτά, τα περισσότερα αυτά χρήματα, τα, τους επιπλέον αυτούς πόρους, κοιτώντας ε, τις εκθέσεις του θεωρητικού συνεδρίου, σε ό,τι αφορά τη συνοχή, σε ό,τι αφορά την Γεωργία. Χθες ε, κοιτάξαμε ε, μια έκθεση του Εθνικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά 18 δισεκατομμύρια για την ε, βασική επιδοτήση των καθεστών επιδοτήσεων στι Γεωργού. Θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους ε, της Επιτροπής να δουν κατάματα την αλήθεια, να κοιτάξουν και να διαβάσουν τις εκθέσεις αυτές, γιατί με τα χρήματα δεν πετύχαμε πάντα αυτό που θα θέλαμε να πετύχουμε. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα και να σας προειδοποιήσω να μην κάνουμε μια έννοια συζήτηση. Υπάρχουν επαρκή πόροι και όλοι θα πρέπει να εργαστούμε για να τους ε, δαπανίσουμε πιο στοχευμένα. Με μεγαλύτερη απόδοση στην γεωργική πολιτική, 10% των ε, μεγαλύτερων εταιριών παίρνουν 90% των πόρων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι όλο και πιο πολλοί άνθρωποι φαίνεται να αγωνίζονται για πιο πολλούς πόρους. Το θέμα είναι πώς διαμορφώνεται η γεωργική πολιτική. Και αν υπάρχει λογική. Να εξετάσουμε λοιπόν βάσει των νομικών κειμένων κατά πόσο έχει νόημα αυτό που κάνουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν μην ε, αρχίσουμε μια αβάσιμη συζήτηση τις, τελευταίες, τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες ε, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ε, πόροι. Θεωρώ ότι έχουμε αρκετά στοιχεία στη διάθεσή μας και στη συνοχή. Έχουμε και μια ενδιαφέρουσα έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης για το ποιο είναι η πιο επιτυχής ε, χώρα. Τσεχία. Η πιο χαμηλή ενεργεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3%. 5% είναι η επόμενη χώρα, η Πολωνία. Δεν έχουμε εδώ και τριτοκοσμικές χώρες στην Ένωση. Οι δύο αυτές χώρες από τότε που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία. Αυτό ήταν ο στόχο ε, των πόρων που δαπανήθηκαν Α μην υποκρινόμαστε λοιπόν ότι δεν έχει γίνει τίποτα, ότι δεν καταφέρνουμε και ότι έχουμε τεράστια τέτοια προβλήματα. Σα παρακαλώ λοιπόν να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί πιστεύω ότι εν μέρη, τι να σα πω, επιβαρύνουμε και υπερβολικά τι υπηρεσίε για την δαπάνη και την απορρόφηση όλων και περισσότερων πόρων. Γιατί πολύ απλά οι τοπικέ οργανώσει, οι τοπικέ μάλλον υπηρεσίε και οι εθνικές ε, διοίκησει δεν μπορούν να απορροφήσουν πιο πολλού πόρου ε, απαραίτητα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στην ε, Ανατολική Ευρώπη. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν λύνονται όλα με πιο πολλά χρήματα. Και κάτι άλλο που με απογοητεύει σε ό,τι αφορά το συνολικό πακέτο. Αυτό που πάλι μου λείπει είναι μία πραγματική ανάλυση των σημερινών ε, επιτεύγματων. Διάβασα το staff document, δεν είναι όμως ανάλυση των προγραμμάτων αυτή για το πώς, ε, πόσο επιτυχή ήταν τα προγράμματα, τι πέτυχε και τι δεν πέτυχε τόσο πολύ. Πολύ λυπάμαι. Πολύ λυπάμαι γιατί πάλι θεωρώ ότι με τα μάτια δεμένα πάμε να καταθέσουμε νέα προγράμματα. Θα ήταν πάρα πολύ καλό αυτό στη συζήτησή μα. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό που στο πακέτο αξιολογείται, συναξιολογείται μάλλον και το θέμα του κράτους δικαίου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να έχει τη δυνατότητα να συνδέει τους ευρωπαϊκούς πόρους με τις διατάξει του κράτους δικαίου. Γιατί σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε ζητήματα και πολλά θέματα. Δεν τα γνωρίζουμε καν και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν, για παράδειγμα, χρηματοδότηση και παρανομών κομμάτων. Πώς θα το αντιπιστώσουμε αυτό, αν συμβαίνει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ε, ότι ενσωματώνεται το EDF. Και νομίζω ότι καλό θα είναι να συγχρηματοδοτεί και το Κοινοβούλιο εδώ και να έχουμε και εμείς ε, αρμοδιότητα. Και δεν πιστεύω ότι δεν προσπιζόμαστε τις παλιές, την παλιά Ευρώπη, τις παλιές αξίες της Ευρώπης. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις. Υπάρχουν ανακατανομές σε σχέση με τα παλιά προγράμματα. Και δεν θα σα προκαλέσει η έκπληξη ότι εγώ θα ήθελα ακόμα πιο πολλέ ανακατατάξει των πόρων σε σχέση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καλό το πακέτο. Μπορούμε να το βελτιώσουμε βεβαίω. Αλλά θεωρώ ότι είναι ουτοπικό και λάθο να θεωρούμε ότι πρέπει να το κατακρίνουμε Εκβάθρων και να συμπεριφερόμαστε με τρόπο που δεν μας βοηθάει. Σε ό,τι αφορά το Brexit τώρα, η Μεγάλη Βρετανία και η αποχώρηση της μεγάλη Βρετανία. Είναι αντίστοιχη με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση 20 μικρών κρατών. 20. Δεν έχουμε ακόμα κατανοήσει ποια θα είναι η τομή που θα επιφέρει στην ευρωπαϊκή πολιτική η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Όταν ήρθε ο Επίτροπος εδώ στο Κοινοβούλιο, μας είπε ότι ήταν έτοιμος να συμπεριλάβει τις προτάσεις μας στα συμπερίσματά του. Αν δείτε όμως τα περιεχόμενα των δύο εκθέσεων, δεν νομίζω ότι η Κομισιόν έλαβε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό υπόψη τις δικές μας προτάσεις, μάλλον τις αγνόησε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε ενδελεχώς όλα αυτά τα θέματα. Η Κομισιόν έχει δημιουργήσει την αυταπάτη ότι κάποιες χώρες μπορούν να συνεισφέρουν, ε, να εξακολουθούν να συνεισφέρουν λιγότερο και να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που έκαναν μέχρι τώρα δηλαδή. Πολύ ωραία. Αν συνεχίσει κανείς να επιμένει σε αυτή την αυταπάτη, μπορεί να την καταστήσει πραγματικότητα τελικά. Αλλά γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την έκθεση της ομάδας Μόντι για τους ιδίους πόρους. Η Συμφωνία του Παρισιού έχει υπογραφεί, υπάρχει, αλλά δεν έχουμε τα εργαλεία για να την εφαρμόσουμε. Ε, η έκθεση Μόντε όμως, ε, της ομάδας Μόντι, μας δίνει τα εργαλεία για να κάνουμε κάτι. Επίσης, οι φόροι διοξείδου του άνθρακα στα σύνορα. Όταν οι τρίτες χώρες εξάγουν ε, αγαθά και εμείς τα εισάγουμε στην αγορά μας ε, και αυτά τα αγαθά έχουν παραχθεί με μη φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο μπορούμε να επιβάλλουμε φόρους σε αυτά τα προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε την ευκαιρία στις επιχειρήσεις της Ευρώπης να ανταγωνιστούν τις τρίτες επιχειρήσεις επί ίσης Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί αυτά τα εργαλεία δεν τα έχετε συμπεριλάβει στην πρότασή σας Κομισιόν. Φοβάμαι ότι η ομάδα Μόντι δούλεψε ει μάτιν. Η κυρία Γκρέσλερ μίλησε για δίκαιου κανόνε. για την ανάγκη να έχουμε δίκαιους κανόνε. Εγώ είμαι οικονομολόγο, δεν είμαι γεωργό. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε δικαιούς κανόνες. Με βάση τους κανόνες που έχουμε για τη γεωργία, τι κάνουμε. Δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στους γεωργούς στις πλούσιες χώρες και λιγότερες δυνατότητες στους γεωργούς στις φτωχότερες χώρες. Δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε δικαίους κανόνες. τα 555 εκατομμύρια ευρώ, το πλεόνασμα αυτό. Είναι το πρόσχημα που δίδεται ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να πληρώσουν λίγα, λιγότερο του χρόνου. Ένα τέτοιο πλεόνασμα, ένα τέτοιο μάλλον ε, πλεονάζον ποσό δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο να πληρώνουν λιγότερα, λιγότερα τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να επιστρέφουμε λεφτά στα κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη, ε, αν το κάνουμε αυτό, το καταπίστευμα για την Αφρική θα μείνει άδειο. Η επιστροφή αυτού του πλεονάσματος, αυτού του ποσού των 555 εκατομμυρίων ευρώ, οδηγεί σε γραφειοκρατία. όλα τα πλεονάσματα, όλα τα ποσά που περισσεύουν τελικά επιστρέφονται στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι προ το συμφέρον μα. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο να δουλεύει επιτέλου, το οποίο θα είναι χρήσιμο επιτέλου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάουαρτ. Θέλω να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε για απογοήτευση. Όταν η Κομισιόν ανακοίνωσε στις 3 Μαΐου ε, τον προπολογισμό, ε, υπήρχαν τυμπανοκρουσίες για την αύξηση στο νορίζοντα 2020 και για το Εράσμους. Και εγώ ε, ήμουν υπέρ γιατί ήθελα τις αυξήσεις αυτά τα προγράμματα από τη στιγμή που ανέλαβα το αξίωμά μου. Ήμουν υπέρ αυτών των αυξήσεων. Αλλά πρέπει να δείτε ότι αν η Κομισιόν ήξερε ποιο είναι το πλαίσιο αυτών των αυξήσεων τον Ιανουάριο, γιατί τι έχουν περάσει, τέσσερις μήνες για, τον προπολογισμό, για έναν προπολογισμό που θα είναι για μια εφταετία. Αν ήξερε το πλαίσιο αυτό, γιατί θα έπρεπε να έχει κάποιες ιδέες τότε, γιατί ο πρόεδρος της Κομισιόν έλεγε ότι τα προγράμματα αυτά θα τριπλασιάσουν τα κονδύλια τους. Γιατί ήρθε ο κύριο Έτιγκερ στην Επιτροπή Προπολογισμού και μίλησε για διπλασιασμό των κονδυλίων αυτών των προγραμμάτων. Γιατί τελικά οι αυξήσει είναι μόνο ε, ύψους 50% αν πιστέψουμε τα νούμερα. Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν διαχείριζεστε σωστά τις προσδοκίες μας. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Τότε γιατί το κάνετε, γιατί λειτουργείτε έτσι. Επίσης, μέσα στον απλοϊκό μου κόσμο, πέρασαν δύο χρόνια από τη στιγμή που αποφάσισε ανοήτως πώς το Ηνωμένο Βασίλειο να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είχατε αρκετό χρόνο για να δείτε τις λεπτομέρειες, για να καταλάβετε τις επιπτώσεις για το επόμενο πουδουπού. Λογικό θα ήταν να υποθέσουμε ότι εμείς εδώ οι πολιτικοί θα έρθουμε εδώ και θα σας κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Θα πρέπει να το περιμένετε. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι λογικό η Κομισιό να λέει «Α, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν τα είχαμε σκεφτεί, δεν φανταζόμασταν θα γίνουν όλα αυτά». Ε, σα δώσαμε κάποια προσεγγιστικά νούμερα κτλ. κτλ. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι είναι αφελές. Μα λέτε παραμύθια εδώ πέρα. Ή αυτό, ή υπάρχει κάποια ανικανότητα από μέρους σας και μας, ή μας κρύβεται κάτι. Ούτως ή άλλως είναι απαράδεκτο. Επίσης, οι περιορισμοί στο Ταμείο για την Νεολαία είναι πολύ προβληματική. Επίσης δεν αναφέρεται πουθενά η εγγύηση για τα παιδιά. Ήταν ένα πρόγραμμα που υπήρχε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Τίποτα, εξαφανίστηκε αυτό, κρίμα είναι. Επίσης, το Ταμείο για τη μετάβαση ε, από μια οικονομία του άνθρακα σε κάτι καινούριο. Εάν μας ενδιαφέρουν τα κλιματικά θέματα, θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Εάν θέλετε ένα κακό μοντέλο του πώς να μην το κάνετε, ας πούμε, κοιτάξτε τι έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα δείτε, ας πούμε, θα σας πω εγώ τότε για ανθρώπινη μετάβαση. Αξιοπρεπή, ας πούμε, μετάβαση. Βλέπω αυτό το ωραίο έγγραφο, πολύ ωραίο μοιάζει κτλ. Αλλά δεν υπάρχει καμιά λογική για αυτές τις αποφάσεις ή για κάποιες από αυτές τις αποφάσεις. Όταν το Κοινοβούλιο είχε πει ότι υπάρχει ανάγκη για την κλιματική χρηματοδότηση ύψου 30%, στην πραγματικότητα είχαμε, μας δόθηκε δέσμευση 25%. Και στην τελευταία συνεδρίαση, ξέρετε πρώτα πολύ καλά, ότι ακόμα και αυτό το νούμερο αμφισβητήθηκε. Τελικά Ποια είναι η λογική αυτού του 25% αντί για το 30% που είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στο Ταμείο Life, ε, εντάξει, υπάρχει αύξηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αύξηση που χρειαζόμαστε ε, για να υπάρξουν οι δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Ε, υπάρχουν λόγια απογοήτευσης δηλαδή και θα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα για να το βελτιώσουμε αυτό το, αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, και να πω και δύο λόγια για τις επιπτώσεις του Brexit. Ε, είπαμε ότι πρέπει να ξαναδούμε τα νούμερα. Εγώ πιστεύω και νομίζω ότι του επόμενου μήνε θα φανεί ακόμα περισσότερο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο τελικά θα καταλήξει να συνεισφέρει να χρηματοδοτήσει κάποια προγράμματα. Ο Εγώ ζήτησα ε, από τον αρμόδιο υπουργό επίσης κάποιες διευκρινήσεις για τις επιπτώσεις του Brexit ε, στο πρόγραμμα Εράσμους. Δεν έχω λάβει καμία απάντηση, δεν σας, σας ε, θα σε εκπλήξει. Πάντως είμαι σίγουρος ότι από, η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι μεγαλύτερη από αυτά που λέει τώρα. Επίσης, τι θα γίνει και με την Ορβηγία. Εάν η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πολύ μεγαλύτερη, τότε καλό είναι να ξέρουμε με ε, απόλυτη σαφήνεια τι θα συνεισφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο και τι θα πάρει ε, σε ανταμοιβή για αυτή τη συνεισφορά, σε αντάλλαγμα για αυτή τη συνεισφορά, ούτως ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Γουαρία Θαβάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν, την κυρία Καλβίνιο, η οποία ήρθε τελικά και μας έδωσε κάποια στοιχεία, του τουλάχιστον κάποιες εξηγήσεις για το πώς δούλεψε η Κομισιόν και κατέληξε αυτά τα νούμερα. Καταλαβαίνω αυτά που είπε η κυρία Καλφίνιο. Είπε ότι έχουμε ένα νέο προπολογισμό, μια νέα στρατηγική, μια νέα εστίαση και τελικά είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε συγκρίσεις. Αλλά εδώ συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, με τον κύριο Χάουαρντ. Τότε, αφού δεν γίνονται οι συγκρίσει, γιατί ο κύριο Γιούνκερ και ο κύριο Έτιγκερ, α πούμε ο κύριο Έτιγκερ, θα φτάσουμε στο 1,11 ή στο 1,9 ας πούμε του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Γιατί τα έλεγε αυτά. Τελικά, στην πραγματικότητα τα νούμερα δεν άλλαξε. Είναι αυτά που πάντα ήθελε το Συμβούλιο. Το ίδιο και με τις συγκρίσεις. Ο ίδιος ο Επίτροπος, η ίδια η Κομισιόν. Μίλαγε για 5% ε, περικοπές 5% ή αύξηση 100%. Τι είναι αυτά. σε τι βασιστήκατε για να φτάσετε σε αυτά τα νούμερα. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις πολλών, τύπων. Και τελικά ο καθένας συγκρίνει τα νούμερα με τέτοιο τρόπο τόσο ώστε να αποδείξει ότι το επιχείρημά του είναι σωστό. Τουλάχιστον όμως να συμφωνήσουμε ότι θα χρησιμοποιούμε μία ενιαία μέθοδο όλοι μας. Αν ασπίσουμε, αν ε, συγκρίνουμε πού παλιό και πού καινούριο, τι θα κάνουμε. Τουλάχιστον να, να πούμε, θα βάλουμε το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα ή έξω. Αλλά και στι δύο περιπτώσει να κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή, α πούμε, αν συγκρίνουμε πού, πού, παλιό και καινούριο, α πούμε, να βγάλουμε το Ηνωμένο Βασίλειο, α πούμε. Να μιλήσουμε με σταθερέ τιμέ ή με τρέχουσε τιμέ. Όμω να έχουμε ένα ενιαίο τρόπο. Ή θα συγκρίνουμε παλιό και καινούριο πού με τρέχουσε τιμέ ή με σταθερέ τιμέ να μην αλλάζουμε, ας πούμε, κριτήριο ανάλογα με το πρόγραμμα. Επίσης, κάτι άλλο. Παρότι είναι σωστό το να συγκρίνουμε με τρέχουσες τιμές, δεν νομίζω ότι δίνει μια πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει. Γιατί αν συγκρίνουμε τις τιμές του 2014 με τις τιμές του 2027, δεν έχει καμία σχέση. Επίση, όταν λέμε ότι θα αυξήσουμε τι οροφέ κατά 10%, δεν είναι το ίδιο να μιλάμε με τρέχουσε τιμέ ή με σταθερέ τιμέ. Δηλαδή, το να συγκρίνουμε, ας πούμε, με τρέχουσες τιμές από μία χρονιά στην άλλη μπορεί να περάσει, αλλά να συγκρίνουμε τις τιμές του 2014 με τις τιμές του 2027 δεν έχει κανένα νόημα. Και ένα τελευταίο σχόλιο θέλω να κάνω και μετά μια τελευταία ερώτηση. Καταρχάς, ένα σχόλιο για την πρόταση εν γέννη. Ο κ. Γιούνκερ, όταν έκανε τη γενική παρουσίαση στην Ολομέλεια, είπε, αν καταφέρουμε να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες της Ένωσης, δεν θυμάμαι ότι θα χρειαστούμε το 2 ή το 3 του ΑΕΠ, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο. Εγώ δεν πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν θα φτάσει στο 2% του ΕΠ ή στο 3% του ΕΠ. Αλλά από αυτό μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που βλέπουμε τώρα, η διαφορά είναι τερατώδης. Θέλουμε, υποτίθεται, μια νέα Ευρώπη. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις. Θέλουμε νέες αρμοδιότητες, κοινέ κτλ. Αν τα θέλουμε όλα αυτά, τι κάνουμε στην πραγματικότητα. Προσπαθούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά πώς, τετραγωνίζοντας τον κύκλο. Δεν νομίζω όμω ότι η Κομισιόν πρέπει να κάνει αυτό ή δεν πρέπει να κάνει μόνο αυτό. Εγώ ήλπιζα κάτι περισσότερο φιλόδοξο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω πάρα πολλέ ερωτήσει. Γιατί τελικά έχουμε κάποια προσεγγιστικά νούμερα, πολύ γενικά, κάποιε γενικέ εξηγήσει, αλλά υπάρχουν προγράμματα τα οποία είναι σχετικά καινούρια, όπω το EU Invest Fund, πάνω στα οποία θα ήθελα περισσότερε πληροφορίε. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα όπου από κάτω από το πρόγραμμα βάζεται τμήμα αυτών των ε, πιστώσεων ή χρημάτων θα χρησιμοποιηθούν με βάση το EU Invest Fund. Αυτό λοιπόν το βάλατε στην ε, γραμμή προπολογισμού του EU Invest Fund ή θα πρέπει να τα αθροίσουμε ας πούμε. Τα νούμερα θα αλλάξουν πάρα πολύ. Στο κόσμο υπάρχει ένα τμήμα των ποσών, των χρημάτων ε, που αφορά τις νέες ευρωπαϊκές επενδύσεις. Μπαίνουν αυτά τα λεφτά στον προπολογισμό ή όχι. Στο νέο κοινωνικό ταμείο ας πούμε. Λέτε ότι με βάση την ε, διαδικασία πλούστευσης και τη γραμμή απλούστευσης θα βάλουμε όλα τα ποσά που πριν υπήρχαν ε, ε, για κοινωνικά θέματα σε αυτό το ταμείο. Όμως εξαφανίζονται διάφορα προγράμματα ή θα, ή θα, ή θα εξακολουθήσει να υπάρχει ας πούμε, η θα η θα εξακολουθησει να υπαρχει ας πουμε εγγυηση για την νεολαία. Θα κρατήσετε ένα πρόγραμμα όπως αυτό της εγγύησης για την νεολαία ε, τη στιγμή που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανεργία ή όχι. Επίσης, τμήμα των προσφύγων είναι μετανάστες. Ε, ένα τμήμα της χρηματοδότησης που θα χρειαστεί θα το καλύψουμε από το νέο κοινωνικό ταμείο. Ναι ή όχι. Θέλω εξηγήσει λοιπόν για αυτό το νέο κοινωνικό ταμείο. Γιατί αν έχουμε τόσα κοινωνικά προβλήματα, υποτίθεται δίνουμε έμφαση σε αυτά τα θέματα και μειώνουμε τα, τα ποσά, δεν έχει νόημα. Επίση, για την Ευρωζώνη, ποια είναι τα, τα κονδύλια, πώ θα ε, λειτουργήσει, ποιε μεταρρυθμίσει θα έχουμε στην Ευρωζώνη. Επίση, ε, οικονομικά εργαλεία, ε, χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Εδώ έχουμε κάποια νούμερα και λίγε εξηγήσει. Θέλω περισσότερε λεπτομέρειε. Από όλα όσα που μα παρουσιάσατε για αυτά τα νούμερα, τι ποσοστό θα πάει στα χρηματοπιστωτικά μέσα. Έχετε κάνει κάποιο υπολογισμό έχει κάποια νούμερα η Κομισιόν. Γιατί άλλε είναι οι εγγυήσει, άλλο είναι τα δάνεια. Τι ποσά μιλάμε για την κάθε κατηγορία, α πούμε. Δεν έχουμε ε, καθόλου πληροφορίε. Επίση, ε, ο κοινωνικό πυλώνα. Έχουμε τη δήλωση του Γκέτεμπουργκ. Τελικά, ε, αυτό που υπάρχει στο σημερινό κοινωνικό πυλώνα είναι κατώτερο από αυτό που υπήρχε παλιότερα. Επομένω, σε τι χρησιμεύσε η δήλωση του Γκέτεμπουργκ, τι άλλαξε. Αυτά είναι κάποια προκαταρτικά και δειγματοληπτικά ας πούμε, στοιχεία που σας δίνω. Έχω πάρα πολλά ακόμα να πω. Χρυστοφόρου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η πιο σοβαρή και κρίσιμη υπόθεση που έχει ενώπιον του σήμερα μέχρι τι ευρωεκλογέ στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο που ουσιαστικά είναι το πώ χτίζουμε την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Ποια Ευρώπη χτίζουμε. Θα συμφωνήσω πλήρω και απόλυτα με τον αγαπητό συνάδελφο τον κ. Μανουέλ Φερνάντε σε όλε τι επισημάνσει καθώ και με αρκετού συναδέλφου. Και αυτό που έχω να πω σήμερα είναι ότι μέσα από τι συγκεκριμένε περικοπέ, όσοι φιλότιμη προσπάθεια και να έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, είναι ξεκάθαρο ότι μιλούμε για περικοπέ δεν ήρθαν αυξήσει, ήρθαν περικοπέ και μάλιστα στο πιο ευαίσθητο σημείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η υπερτουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνοχή, που έχουν να κάνουν με την αλληλεγγύη. Μα η Ευρώπη που θέλουμε και επιδιώκουμε, που είναι η σωστή Ευρώπη και την επιδιώκουμε μέσα από το πολιετέ δημοσιονομικών πλαίσιων που έφτιαξαν οι αγαπητοί συνάδελφοι εισηγητέ και σκιώδει, που είναι μια Ευρώπη που θα ανταποκρίνεται στι προκλήσει τη νέα εποχή. Ευρώπη χωρί ενισχυμένη κοινωνική συνοχή χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς στήριξη τη υπαίθρου, της γεωργίας, χωρίς ενισχυμένα μέτρα που θα δημιουργούν μια κοινωνική Ευρώπη με μια κοινωνική πολιτική, δεν είναι η Ευρώπη που επιδιώκουμε και η Ευρώπη που θέλουμε. Άλλωστε θεωρώ ότι με αυτέ τι συζητήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιστρατεύεται την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον πρόεδρό τη, τον, τον κύριο Γιούγκερ, ο οποίο ουσιαστικά στι ομιλίε του για το μέλλον τη Ευρώπη μα μίλησε για την Ευρώπη ακριβώ που θα ανταποκρίνεται στι προσδοκίε των πολιτών και όχι στι προσδοκίες των τεχνοκρατών. Επιτέλου πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι λαμβάνουν τι αποφάσει για το μέλλον τη Ευρώπη και για την Ευρώπη που θέλουμε και διεκδικούμε. Οι τεχνοκράτε ή ή οι λαοί με του πολιτικού. Και ένα πολύ σημαντικό. Πολλέ φορέ συζητούμε εδώ μέσα για τον ευρωσκεπτικισμό, για την αύξηση και την άνοδο κινημάτων ενάντια στην Ευρώπη, ακραίων κινημάτων με αυτόν το δημοσιονομικό πλαίσιο που μας προτείνεται και τις περικοπές οι Ευρωπαίοι θα αγκαλιάσουν το νέο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο ή θα αυξήσουμε ακόμα περισσότερο αυτόν που τάχατες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον ευρωσκεπτικισμό και την αποστροφή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ότι έφυγε η Μεγάλη Βρετανία είναι σεβαστό. Αλλά εδώ είναι που πρέπει να αποδείξουμε ότι με τη φυγή τη Μεγάλη Βρετανία η Ευρώπη συνεχίζει ενισχυμένη και δυνατή αυξάνοντας αυτές τις πολιτικές που είναι για μια Ευρώπη κοινωνική, μια Ευρώπη που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα των πολιτών, μια Ευρώπη που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αγροτών της περιφέρειας. Και ένα τελευταίο κύριε Πρόεδρε, ένα τελευταίο. Θα συμφωνήσω κι εγώ με κάποιους συναδέλφους όσον αφορά την Τουρκία. Εδώ είμαστε η Ευρώπη της δημοκρατίας. Εάν μια χώρα όπως η Τουρκία κατάργησε όλους τους κανόνες του δικαίου, καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα, προσβάλλει και προκαλεί χώρε όπω την Ελλάδα και την Κύπρο καθημερινά και ουσιαστικά πλήττει τα συμφέροντα ευρωπαϊκών χωρών ακόμα και τη Ιταλία. Μα είναι δυνατόν, παρά το ότι η Ευρωπαϊκή, εμεί ω Επιτροπή Προπολογισμού περικόψαμε 200 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ορθό να πάει εισήγηση από την Επιτροπή Προπολογισμού όταν δεν εφαρμόζονται αυτέ οι αρχέ να παγώσουν τα προενταξιακά κονδύλια τη Τουρκία και τη οποιασδήποτε χώρα έχει ανάλογη συμπεριφορά. Εδώ παίρνουμε μέτρα κυρώσεων ακόμα και για χώρε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μα φοβίζει να πάρουμε μέτρα για μια χώρα που δεν εφαρμόζει τίποτα και περιφρονεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά θα κάνουμε και εξοικονόμηση στου προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Κύριε Μαλέτιτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι χωρίς λεπτομερείς συγκριτικούς πίνακες δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς τι υποστηρίζουμε και τι όχι από την πρόταση της Κομισιόν. Στην βάση των διαθέσιμων πληροφοριών, ωστόσο, εγώ αναγνωρίζω ότι έχω σημαντικό πρόβλημα με τα προτινόμενα μηνύματα και πολιτικούς στόχους από την πρόταση που έχουμε επιτάπητος δηλαδή. Και θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν εξετάζουμε τον έρασμο, όλοι συμφωνήσαμε ότι ο έρασμος πρέπει να αυξηθεί. Είναι σημαντικό πρόγραμμα κινητικότητας, ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και όχι μόνο μεταξύ νέων ανθρώπων, αλλά και καθηγητών κλπ. Απ' την άλλη μεριά, για ιστερούσες περιφέρειες και για λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, εάν ταυτόχρονα δεν επενδύσουν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καλής ποιότητας να επενδύσουν σε παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Αν περικόψουμε αυτές τις επενδύσεις σε αυτές τις περιφέρειες, τότε η κινητικότητα θα γίνει στην ουσία μόνιμη μετανάστευση. Θα θέσουμε έτσι λοιπόν σε μεγάλο κίνδυνο αυτές τις ιστερούσες περιφέρειες, διότι θα τους λείψει το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα πάει να εγκατασταθεί σε πιο ανεπτυγμένες χώρες και το μήνυμα που δίνουμε με την πρόταση αυτή είναι επικίνδυνο. Αφού πρόκειται για περίοδο επταετίας και μπορεί να αλλάξει σε βάθος το ευρωπαϊκό μέλλον. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την Εννοητική Αριστερά. Τέσσερα πράγματα. Πρώτο. Η ομάδα μου συμφωνεί με το γεγονό, με την ιδέα μάλλον ότι χρειάζεται, υπάρχει ένα καθήκον αλήθεια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για του αριθμού, Πρέπει να μπορούν να αξιολογηθούν οι πολιτικές που έχουν ήδη διεξαχθεί τώρα. Μετά πρέπει να μπορούμε να επιλέξουμε κλίμακες και χρειαζόμαστε τα σχετικά νούμερα. Και επίσης, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα ζήτημα δυσπιστίας που φαίνεται στην ε, συζήτηση και λένε και στα γαλλικά ότι όταν υπάρχει ασάφεια εμφανίζεται ο λύκος και τρώει τα προβατάκια. Εγώ θέλω λοιπόν να πω πρώτον για τον όγκο του προπολογισμού. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο προπολογισμό για ένα απλό λόγο. Μιλούν πολλοί για το Brexit, για την μείωση του αριθμού των χωρών που είναι καθαρή εισφορής. Όμως, εγώ θεωρώ ότι κυρίως πρέπει να κυριαρχήσουν οι ανάγκες του κόσμου, του κοινού, των πληθυσμών. Κάτι που δεν αποκλείει στο εσωτερικό του προϋπολογισμού αυτού να είναι ανάγκη να γίνει κάποιος αναπροσανατολισμός των πολιτικών όπως της κοινή αγροτικής πολιτικής αλλά και κάποιων άλλων. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο οικολογικό, κοινωνικό και δημοκρατικό πρόσωπο. Για τους προσανατολισμούς που μας δίνονται σήμερα, εκεί συνυπογράφω τα όσα λέχθηκαν, όμως είμαστε αντίθετες με τη μείωση του προϋπολογισμού για την αγροτική πολιτική. Είμαστε αντίθετες με τη μείωση του προϋπολογισμού της συνοχής. Και έχουμε και κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τα στοιχεία που μας δίνονται σε ό,τι αφορά την νεότητα. Εξ αντιθέτου, ανησυχούμε και για οποιαδήποτε αύξηση του προϋπολογισμού. Αύξηση δηλαδή για το προϋπολογισμό της άμυνας, καθώς και του Frontex, που δείχνουν μια Ευρώπη που σκέφτεται περισσότερο την ασφάλεια. Θέλω να μιλήσω ακόμα και για τους νέους πόρους. Υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα σε αυτό που λένε «Α, πρέπει να μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις των πολιτικών». Αλλά από την άλλη μεριά χρειαζόμαστε νέους πόρους. Δεν μας αρέσει το γεγονός ότι τελικώς δεν προωθείται ο φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Κάτι το οποίο απασχολεί το κοινό. Από τη μια μεριά μειώνουμε τα κονδύλια της αλληλεγγύης και από την άλλη υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν φορολογούνται. Ούτε μας αρέσει το σενάριο για τον ε, φόρο που επιβάλλεται σε ενέργειες που παράγουν για του θερμοκηπίου. Τέλος, για την γενικότερη ε, δόμηση του προϋπολογισμού, θεωρούμε ότι για να μειωθούν οι λαϊκισμοί και οι εθνικισμοί, πρέπει να δοθεί μια νέα κοινωνική όθηση στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, και επομένω, οι προσανατολισμοί του προπολογισμού για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να, και, να τοποθετηθώ προσωπικά αυτή την, σε αυτή τη φάση, πριν δώσω το λόγο πάλι στους συζήτητες. Πρώτον, χαιρετίζω το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι δεν είναι εύκολο να φτιαχτεί προπολογισμό για τα χρόνια 2021 έω 2027, όταν ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το ερώτημα για ποια Ευρώπη μιλούμε. Ποιο είναι το ευρωπαϊκό project. Τούτου λεχθέντος ερώτηση, κυρία Καλβίνιο, για την συνοχή. Διότι Υπάρχει ταμείο συνοχή το οποίο δεν περνά από τον προπολογισμό. Νορβηγία και Ελβετία συνεισφέρουν τα έχει πει ο κύριος Μόντι και η ομάδα υψηλού επίπεδου, ότι δηλαδή η κοινή αγορά έχει μια αξία και, και η απόδειξη είναι ότι και η Νορβηγία και η Ελβετία πληρώνουν εισφορές για να συμμετέχουν στην κοινή αγορά, στην ενή αγορά. Οι πόροι που χορηγούνται από Νορβηγία και ε, Ελβετία δεν μπαίνουν στον προπολογισμό. Εάν η Μεγάλη Βρετανία στη διάρκεια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων δεχθεί να καταθέσει συνεισφορά και αυτή για να μπορεί να παραμείνει εντός της ενιαίας αγοράς, πού θα εμφανίζονται τα έσοδα αυτά, κυρία Καλβίνιο. Δηλαδή, θα δούμε για άλλη μια φορά ένα είδος απόκρισης. Πού θα μπουν, θα μπουν στον προϋπολογισμό. Όταν μιλούμε για συνοχή, πού είναι τα εκατομμύρια πληρών Ελβετία και Νορβηγία. Είπατε επίσης για να προχωρήσει ο προϋπολογισμός, διότι εδώ συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε δεν μιλούμε για να δαπανίσουμε περισσότερα ως αυτού σκοπό. Χρειαζόμαστε δαπάνες συνολικά. Χθες είχα προσκληθεί από την ομάδα της οποίας ηγείται η κυρία Χολμάιρ για, το, για θέματα του διαστήματος. Βεβαίω το διάστημα δεν γνωρίζει σύνορα και εκεί έχουμε Κοπέρνικο, έχουμε Γαλιλαίο, έχουμε και άλλες εφαρμογές που έχουν σημαντικέ επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών και μάλιστα θέλουμε να γίνουν και πιο γνωστές. Πάντοτε υπάρχουν όμως δαπάνες στο εθνικό επίπεδο για το διάστημα. Έχετε προχωρήσει σε διάλογο με τις χώρες μέλη για να ρωτήσετε τι ακριβώς χρειάζονται. Αντί να δαπανάτε τα χρήματα, ας πούμε, στο εθνικό επίπεδο, δεν είναι καλύτερα να δαπανηθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Να δώσω τώρα το λόγο στους εισηγητές πάλι με την αντίθετη ε, φορά που χρησιμοποίησαμε προηγουμένως και θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Ντεπρέ. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πολλά σχόλια να κάνω. Αναμένω τα έγγραφα με τα συγκριτικά δεδομένα για να μπορούμε να δούμε τις αλλαγές που γίνονται Νομίζω ότι ένα ουσιώδες μέρος της εργασίας μας θα μπορέσει να γίνει με σωστό τρόπο μόνο όταν θα έχουμε και συγκεκριμένες πληροφορίε για το περιεχόμενο των νέων προγραμμάτων. Πρόκειται για δύο θεμελιώδη στοιχεία. Πρώτον, οι αριθμοί που θα μας επιτρέπουν πραγματική συγκρισιμότητα και δεύτερο, συζήτηση ουσίας για το περιεχόμενο των προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Λεβαντόφσκι. Νομίζω ότι εδώ βλέπουμε μία μικρή απόκληση. Στο τελευταίο προπολογισμό πριν από ήταν και 27 και όχι 28 χώρες, γιατί η Κροατία θα προστίθεται αργότερα το 2014. Και πάλι ε, αναμέναμε συγκρίσιμα στοιχεία σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ολμπρίχτ. Νομίζω ότι περιμέναμε να εργαστούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του Συμβουλίου. Θα θέλαμε να είμαστε σε νέο μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά για να είμαστε μαζί θα πρέπει να έχουμε όλα τα αριθμητικά στοιχεία στη διάθεσή μας και θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Αν δεν κατανοήσουμε τα αριθμητικά στοιχεία, δεν προκαλεί αυτό φυσικά έκπληξη για τους πολιτικούς, αλλά όταν και οι εμπειρογνώμονες που έρχονται ερμηνεύουν τα εθνικά στοιχεία με εντελώ διαφορετικούς τρόπους, ε, μα κάτι πάει στραβά στην περίπτωση αυτή. Και γι' αυτό λοιπόν, από πολιτικής άποψης, Δίκιο έχει η κυρία Γκρέσλε για τη συνοχή, αλλά η περικοπή κατά 45% της, ε, της ε, συνοχής πολιτικώς θα προκαλέσει έκπληξη, έκρηξη συγγνώμη, δεν μιλάμε για μείον 15%, μιλάμε για μείον 45%. Μιλάμε για έκρηξη σε ό,τι αφορά το κόστος, σε ό,τι αφορά τις τιμές. Άρα, και εγώ αναμένω απάντηση στο ερώτημα αυτό. Τι θα γίνει αν δεν υπάρχουν ε, ήδη πόροι που τώρα συγκαταλέγονται στους πόρους. Τι θα κάνουμε, θα περιορίσουμε, θα μειώσουμε τον προπολογισμό αν δεν γίνουν αποδεχτές αυτές οι διδάξεις. Αυτό είναι το εκκρεμές ακόμα ερώτημα. Αν δεν υπάρχει ήδη πόρη, δεν θα υπάρξει και πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. το Τωμά. Μάλιστα. Ευχαριστώ την κυρία Καλβίνια για τις διευκρινήσεις αυτές. Ωστόσο, αν ε, θέλετε σεβασμό, θα πρέπει να δείξει σεβασμό και η Επιτροπή προ το Κοινοβούλιο. Και έχω τι αμφιβολίε μου. Να σα δώσω το εξή ε, παράδειγμα. Ο Επιτροπό ανακοίνωσε σε ό,τι αφορά τον Ορίζοντα 2020 αύξηση, όχι διπλασιασμό ωστόσο. Σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή, 10, μείωση μάλλον, και σε ό,τι αφορά το Εύση είναι 49. Βλέπουμε λοιπόν η πολιτική των να, να μεταμορφώνεται σε μία ε, οικονομικό ουσιαστικά μέσο, το οποίο φυσικά δεν είναι το ίδιο. Πρόκειται για ένα χειρισμό λοιπόν και μετατρέπονται τα ανώφλια κατά 0,9% σε ό,τι ε, ε, τον Εράσμους ε, το 79% το 79% δεν αποτελεί διπλασιασμό. Άρα, κοιτάξτε, εγώ να επιδείξω σεβασμό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να λάβει τον αντίστοιχο σεβασμό και το Κοινοβούλιο. Ενδεχομένω να μην στέκουν όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία που σα ανέφερα. Αν ισχύει όμω κάτι τέτοιο, υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη, γιατί αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε επί των αριθμητικών στοιχείων Εμεί, στο ψηφισμά μα θα βάλουμε τα δικά μα αριθμητικά στοιχεία, Προφανώ. Και θα ξεσπάσει η μάχη. Και αυτό προφανώ είναι απευκταίο. Κανεί δεν το επισημεί αυτό. Και αυτό θα πρέπει να γίνει εν πάσα συντομία. Γιατί η προθεσμία, νομίζω, για την κατάθεση του ψηφίσματο είναι Δευτέρα. Δεν έχουμε ούτε καν μια εβδομάδα. Λιγότερο από μια εβδομάδα. Είτε λοιπόν θα βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε πραγματικά την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, όπως είπε και η κυρία Καρδιά Σαμπάλ πριν από λίγο, επί της μεθοδολογίας. Μία μεθοδολογία η οποία θα ισχύει για όλο το πλαίσιο. Μπορεί να υπάρχουν και δύο μεθοδολογίες, να υπάρχουν πίνακες, αλλά σε κάθε περίπτωση να μιλάμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Να μην επιλέγει ο καθένας ό,τι μεθοδολογία επιθυμεί σε ό,τι αφορά την επίκριση του συστήματος και αυτό τώρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρώ ότι καταπηγόντως θα πρέπει να μην αντιδράσουμε υπερβολικά, αλλά να συμφωνήσουμε επί των αριθμητικών στοιχείων. Ιδάλω, έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου. Πώ θα πετύχουμε συμφωνία με του όρου αυτού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βιαστούμε μέσα στι επόμενε εβδομάδε, προκειμένου και το ψήφισμα να αναφέρει αριθμητικά στοιχεία από τα οποία συμφωνούμε. Αλλιώ, επαναλαμβάνω, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά που ερμηνεύουμε εμεί ω Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρο. Μάλιστα, δούμε λοιπόν ε, α ε, διατηρήσουμε την ψυχραιμία μα, να μην ξεκινήσουμε αντιπαλότητε και διαμάχε για τα αριθμητικά στοιχεία. Προφανώ χρειαζόμαστε μια φιλοδοξία. Η κυρία Καλβίνιο ενδεχομένω θα ήθελε να πάρει το λόγο για να κάνει κάποια συμπεριφηματικά σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τα μέλη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για τα σχόλια τους, τα οποία θεωρώ ότι είναι πραγματικά ωφέλιμα και επικοδομητικά για τη μελλοντική συνεργασία μας. Τρία σημεία, εν συντομία, επιτρέψτε μου να αναφέρω. Καταρχάς, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε σε ό,τι αφορά τα διάφορα θέματα που αναφέρθηκαν. Νομίζω ότι προφανώ θα πρέπει να γίνει ένα τεχνικό σεμινάριο, ένα εργαστήριο και με χαρά θα έλθω να συζητήσουμε τι λεπτομέρειε αυτέ. Απλά να αναφέρω ότι στο πακέτο που δημοσίευσαμε έχουμε την ανακοίνωση και έχουμε και κάποια σχέδια που εξηγούν πώ προέκυψαν τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία δημοσιεύσαμε και τα οποία ανακοίνωσε ο επίτροπο και υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος των προγραμμάτων και των ε, κονδυλίων ανά πρόγραμμα. Να προσπαθήσουμε επίσης να κοιτάξουμε και τα έγγραφα τα οποία δημοσιεύσαμε στην έκθεση δαπανών. Τα έχει αναλύσει ήδη η κυρία Κρέσλε. Είναι μεγάλη πληθώρα των δεδομένων αυτών και των στοιχείων αυτών και τα έχουμε δημοσιεύσει σε ό,τι αφορά τα διάφορα προγράμματα. Όπως είπε ο κύριος Δεπρέ, επί του παρόντος. Αυτό έχουμε επιτάπητος. Θα πρέπει να περιμένουμε τα, προ... τα τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων. Το πρώτο πακέτο περιμένουμε να δημοσιευτεί στα τέλη του μήνα σε ό,τι αφορά τη συνοχή και τη γεωργία. Πολύ σημαντικό πακέτο και αυτό προφανώς θα αρχίσει να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και ελπίζω μέχρι, 15, μέχρι 12 Ιουνίου να έχουμε ε, το πλήρες πακέτο μπροστά μας. Να σας ε, Βεβαίω ότι επί κάποιων στοιχείων μπορούμε να ξεκινήσουμε ήδη να δουλεύουμε. Για κάποια άλλα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί δεν έχει ολοκληρώσει τη δουλειά του το σώμα των επιτρόπων. Αλλά προφανώ θα επισέλθουμε σε λεπτομέρειε. Δεύτερο σχόλιο. Κάποιοι αναφέρθηκαν στους ιδίους πόρους. Έχουμε κάνει ενδελεχή εργασία και έχουμε και ένα κεφάλαιο για τους ιδίους πόρους στο πακέτο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εξετάσουμε όλες τις εναλλακτικέ ε, λύσεις της ομάδας και της έκθεσης Μόντι και κάποιες επιπλέον. Για παράδειγμα, η συνεισφορά βάση πλαστικού δεν συμπεριλαμβανόταν στην έκθεση Μόντι και υπάρχει και μια ενταλλαχέστατη ανάλυση του τι πιστεύουμε ότι θα λειτουργούσε και τι όχι. Γι' αυτό λοιπόν και απορρίψαμε ε, κάποιες ε, λύσεις, όπως για παράδειγμα αφορούσε ε, για το διοξείδιο του άνθρακα. Ε, να προσθέσω και την ε, ψηφι... έκθεση για την ψηφιοποίηση και για τον φόρο οικονομικών συναλλαγών. Από το 2011, αν δεν κάνω λάθο, είχε προταθεί και θεωρήσαμε ότι δεν ήταν λογικό να το υπολογίσουμε και να το συνυπολογίσουμε ω έσοδο στο άμεσο μέλλον. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι το έχουμε καταλήψει πολιτικά ω ιδέα, αυτή την πρωτοβουλία δηλαδή. Όχι, θέλαμε να υποβάλουμε προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εγκριθούν μέχρι τον επόμενο Μάιο και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο επόμενο πουδουπού. Τρίτον, τρίτο σχολείο, σε ό,τι αφορά τα σχολεία του Προέδρου για τη συνεισφορά α, τρίτων χωρών. Κάποιε συνεισφορέ ε, είναι, είναι πόροι που έχουν ανατεθεί για συγκεκριμένα προγράμματα, Κάποιε είναι διμερεί ε, συνεισφορέ που έχουν συμφωνηθεί διμερώ με τις χώρες και αυτέ δεν περνούν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Αλλά στο μέλλον, εφόσον ε, αν υπάρξει για παράδειγμα συνεισφορά από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα εξαρτηθούν όλα από την φύση της συμφωνίας. Μπορεί να πρόκειται για πόρους που θα ανατεθούν συγκεκριμένα για κάποιο πρόγραμμα, μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο άλλο πλαίσιο. αυτό θα ισχύσει μετά τον Brexit. Δεν θα υπάρχουν πλέον ήδη πόροι από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά αν υπάρξει συμφωνία και βάση των ε, συμφωνιών που έχουμε σήμερα θα έχουμε άλλα έσοδα, άλλα πρόσοδα από τον Εμμανό Βασίλειο στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό που θα περάσουν για το σύνολο του προπολογισμού. Αλλά, επ' να τονίσω και το εξή. Μία από τις προσπάθειες που κάναμε είναι να προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε, να πλουστεύσουμε ε, το γαλαξία που αναφέρεται συνέχεια σε ό,τι αφορά την, ε, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, σε ό,τι αφορά τα άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση στον ευρωπαϊκό προπολογισμό των εργαλείων που σχετίζονται με την Ευρωζώνη, κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να απλοποιήσουμε το συνολικό οικοδόμημα του ευρωπαϊκού προπολογισμού και πιστεύω ότι στο μέλλον Πιο σωστό είναι να μην βγαίνουν πράγματα από τον προπολογισμό, αλλά να υπάρχει ένα πιο αναποιημένο πλαίσιο και να περνάει φυσικά από τον ανάλογο έλεγχο. Σα ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τα αρχικά σας σχόλια. Προφανώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω διευκρινήσεων. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό το συντομότερο δυνατόν και μπορείτε να υπολογίσετε σε εμά. Θα είμαστε όσο πιο δυνατόν επικοδομητικοί στην συζήτηση αυτή. Σα ευχαριστώ. θα τιμήσουμε την Κομισιόν για την προσπάθειά τη να δώσει διευκρινήσει, ούτω ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να, για να βγούμε τέλο πάντων από το αδίέξοδο. Θα πρέπει να σεβαστούμε την ενότητα του προπολογισμού. Είναι μια βασική αρχή. Αλλά, κυρία μου, οι συνεισφορέ που δίνει η Νορβηγία ας πούμε, και η Ελβετία, γιατί δεν περνάνε μέσα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και πάνε κατευθείαν ας πούμε, ε, στο Ταμείο Συνοχή. Τι πράγμα δικαιολογεί αυτό αυτή τη μέθοδο. Μπορείτε να μου πείτε. Ο συνάδελφος προσπαθεί να δει τις λεπτομέρειες. Ε, γιατί εγώ θεωρούσα και μου το επιβεβαίωσε ότι είναι, αυτά βασίζονται σε διακυβερνητικές ε, συμφωνίες. Κάποια από τα, στοιχεία επίσης ε, στο μέλλον θα είναι τμήμα αυτού του μηχανισμού διευκόλυνση τη Ειρήνη. Ε, δεν θα περνάνε μέσα από τον προπολογισμό. Αυτό προσπαθούμε βεβαίω στο, προσπαθούμε στο μέλλον είναι να βάλουμε περισσότερα από αυτά τα στοιχεία μέσα στον προπολογισμό. Αλλά δεν μπορούμε να ε, προδικάσουμε ποια θα είναι η μελλοντική φύση τη ε, μα μας ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο τη στιγμή που δεν έχουμε συμφωνήσει για την, ε, το πώς θα αποχωρήσει. Κοιτάξτε τι θέλω να σας πω. Τα ποσά που πάνε στη συνοχή όλα όσα είναι στον προπολογισμό δεν είναι το 100% των ε, πιστώσεων της ε, συνοχής. Καλό θα ήταν να ξέρουμε κάθε κράτος μέλος που εποφελείται από τη συνοχή, τι παίρνει από τις συνεισφορές που καταβάλει η Νορβηγία και η Ελβετία. Καλό θα ήταν για λόγους ευκρίνειας. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Ε, θα σταματήσουμε τώρα, θα ξαναρχίσουμε στις 2.30 θα κάνουμε μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, της οποίας προεδρεύει η κυρία Γκρέσλερ και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που έχει πρόεδρο τον κύριο Μωράες. Σταματά εδώ η πρώτη μας συνεδρίαση και ξαναρχίζουμε στις 2.30.